propose de prendre place. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας. Bien, je propose tout Προτείνω, εάν συμφωνείτε, να εγκρίνουμε χωρίς τροποποίηση στην ημερήσια διάταξη. Δεν έχετε αντίρρηση. καλά και ευχαριστώ. Μερικές ανακοινώσεις. Διερμηνία έχουμε ως συνήθως πλην του, της Εστωνικής, λετονικής και μαλτέζικης γλώσσας σήμερα. Δεύτερον, 17 ε, Οκτωβρίου από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα έχουμε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την ετήσια συνάντησή μας με την κυρία Ζακλίν Ματή, την την Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος. 3 με 6, 18 του μηνό. Και επίσης θα έχουμε επίσκεψη από μια ομάδα προερχομένη από τη Γερμανία, επισκέπτες από τον Ρηθό Σταυρό. Καλώ ήρθατε, κάπου τώρα μπαίνουν στην αίθουσα. Θα παρακολουθήσουν τις εργασίες μας περίπου και 40 λεπτά. Και τέλος, το σύστημα των ποσοστώσεων, της ανταλλαγής ποσοστώσεων εκπομπής. Έχουμε 700 εκατομμύρια, 698 συγκεκριμένα πιστώσεις ε, ανταλλαγών εκπομπών για την περίοδο στο 2019. Δωρεάν πιστώσεις που υπάγονται στην απολύτευση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θα μας ε, ετοιμάσει γνωμοδότηση μέσα σε περίοδο 6 μηνών. Νέα κυβέρνηση στη Δανία μετά τις εκλογές. Ίντα Χόκεν, σοσιαλίστρια και κόρη του Σβέν Χόκεν, που εγώ προσωπικώς είχα γνωρίσει, αναλαμβάνει υπουργό περιβάλλοντος της υγείας, υπουργό η Άστριτ Κράκ, από το Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα. Η ΔΕ Μάρτιν Λίτεκαρτ αναλαμβάνει εκ μέρους του ε, ριζοσπαστικού κόμματο, ο Υπουργό Αρμόδια για θέματα των καταναλωτών. Η κυρία Χέκ επίσης, ε, συνάδελφος, αναλαμβάνει ε, Υπουργό Περιβάλλοντος στη Σουηδία και τη ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Αυτά για τι ανακοινώσει μας. Στην εμείς διαταξή έχουμε επίση την πρόταση για έγκριση των πρακτικών 23 25 Μαΐου του 2011 και αντίστοιχα Ιουλίου του 2011. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, σας ευχαριστώ πολύ. Εγκρίνονται και τώρα περνάμε στο πρώτο θέμα τη ημερήσια διάταξης, Στρατηγική, διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετεί τον που ε, είναι προς το συμφέρον του πολίτη, στην υπηρεσία του πολίτη και η συγκητής είναι ο κύριος Ταραντουμπέλα, στον οποίο και δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 4 Απριλίου η Επίτροπη υπέβαλε μία ανακοίνωση, εξέδωσε μία ανακοίνωση για τη διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του πολίτη. Εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε, ενώ η αρμόδια επιτροπή είναι Επιτροπή Βιομηχανίας. Το έγγραφο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό, διότι η ίδια Επιτροπή, λίγους μήνες μετά, στις 4 Απριλίου, με μία ακατανόητη η στάση και ίσως και καθαρά σχιζοφρενική και συγγνώμη για τον όρο, διέγραψε το πρόγραμμα ΓΜΕΣ από, το, από την πολιετή χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή στον ε, πολιετή της προϋπολογισμό δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει το ΓΜΕΣ που είναι ένα πολύ βασικό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα σύμφωνα με την Κομισιόν θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη, τα οποία θα πρέπει να διαθέσουν τα κατάλληλα κονδύλια. Δηλαδή 843 εκατομμύρια ετησίως θεωρώ ότι αυτή η επιλογή είναι λανθασμένη και θα πρέπει να αντιταχθούμε διότι θα πρέπει να εκφραστούμε ομόφωνα και το ζητώ από την Επιτροπή, να είμαστε δηλαδή ομόφωνοι έτσι ώστε να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αλλάξει κατεύθυνση και να ταχθεί υπέρ της χρηματοδότησης του ΓΜΕΣ. Εμείς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Επιτροπή αρνήθηκε να χρηματοδοτήσει ένα από τα προγράμματά της και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε επίπεδα λήψης αποφάσεων η Επιτροπή έχει μεγάλη δυσκολία να εγκρίνει επιστημονικά προγράμματα τύπου ΓΜΕΣ. Γιατί θα πρέπει να πω ότι σχεδόν καθημερινά ασχολούμαστε με θέματα υπέρ του περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής. Το ΓΜΕΣ θα μπορούσε να μας βοηθήσει ιδιαίτερα για αυτά τα ζητήματα, διότι παρακολουθεί το περιβάλλον και για θέματα ασφάλειας, ασφάλειας της Ευρώπης, εποπτείας, εποπτείας των ε, συνόρων. Και το λέω και από πλευρά Ιταλών, αλλά και για τους Γάλλους και τους Ισπανούς υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και το ΓΜΕΣ θα μπορούσε να μας βοηθήσει στις σχέσεις μας με τις ε, χώρες της Βορείου Αφρικής. Δηλαδή να επαυξήσει τη συνεργασία στη Μεσόγειο. Θα μας βοηθούσε λοιπόν με αυτή τη χρηματοδότηση που ανέρχεται στα 850 εκατομμύρια κατά μέσο όρο να βοηθήσουμε αυτή την παρακολούθηση και πιστεύω ότι αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να ανακτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή. Ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο συνάδελφος Θαταρέλα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω, πέρα από αυτά που είπε, και τον ε, ρόλο αυτών των υποδομών που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, είναι αναντικατάστατες για την εφαρμογή γενικότερα της ευρωπαϊκής πολιτικής υπέρ του διαστήματος. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και μην ξεχνάμε και το πρόγραμμα ε, Galileo και το Σέζαρ, τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και ένα, το νέο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, που θα μας επιτρέψει να εξοικονομήσουμε κατά 15% σε καύσιμα, γιατί θα εξορθολογήσουμε τις εναέριες διαδρομές και θα αντιμετωπίσουμε και την συμφόρηση των αερολιμένων. Όσον αφορά τις προσγειώσεις, απογειώσεις και τις χρονοθυρίδες. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι απολύτως ε, αναγκαίο κάτι τέτοιο για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα διάφορα προγράμματα δορυφόρους που υπάρχουν στα προγράμματα της Επιτροπής. Θα ήθελα να κινηθούμε και πέραν αυτών που είπε ο κύριος Ταταρέλα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να διακόψουμε τη χρηματοδότηση του ΓΜΕΣ ιδιαίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το ΓΜΕΣ επηρεάζει όλες τις πολιτικές ελέγχου ε, αερίων θερμοκηπίου και αφορά είτε την ε, υπερθέρμανση καθώς και όλες τις ε, πολιτικές διατήρησης των δασών, ιδιαίτερα των τροπικών δασών. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με προγράμματα δορυφόρους που θα πρέπει να υποστηριχθούν. Πρόκειται για μια βασική ευρωπαϊκή υποδομή. Δεν θα πρέπει να ζητούμε χρηματοδότηση των μεμονωμένων κρατών μελών, γιατί πρόκειται για ομαδοποιημένα ευρωπαϊκά προγράμματα και έτσι τα διαχειριζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον λοιπόν πρόκειται για ευρωπαϊκές υποδομές, θα ήθελα να σταθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μπαρόζο στην ανακοίνωσή του προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο όταν μίλησε για την κατάσταση της Ένωσης. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα λέει, και θα ήθελα να ζητήσω τη συμφωνία των συναδέλφων έτσι ώστε να προωθήσουμε μία πιο ενισχυμένη δράση. Εάν μιλάμε για ευρωπαϊκές υποδομές, θα πρέπει να βρούμε και τον κατάλληλο χώρο στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και επειδή διανύουμε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση, αυτές οι υποδομές αποτελούν παράδειγμα χρηματοδότησης, πολιετούς χρηματοδότησης που είναι απολύτως αναγκαία για τη συνέχισή τους γιατί εκεί βασιζόμαστε για να δημιουργήσουμε τη μελλοντική μας, να υποστηρίξουμε τη μελλοντική μας πορεία. Χρειάζεται λοιπόν μία θαραλέα χρηματοδότηση, μία προετοιμασία για το μέλλον μας και μία χρηματοδότηση που θα ήταν αποφασιστική σημασίας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την κρίση στο σύνολό της. Ας δούμε λοιπόν αυτές τις χρηματοδοτήσεις ως ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και ας δείξουμε θάρρος δίνοντας όθηση σε αυτά τα προγράμματα, διότι είναι απολύτως αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε και την τρέχουσα συγκυρία, για να μπορέσουμε να βγούμε ενδεχομένως και από την ε, οικονομική αυτή κρίση. Ε. Σατουάσι, Η κυρία Χάση θέλει το λόγο. Όχι. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ. Εντάχει, απλώς για να σας πω και εγώ ότι υποστηρίζω τους προλαλήσαντες. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος Ήδη το είχαμε συζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη συζήτηση της έκθεσης Γκαρντίνη για την ασφάλεια, την πολιτική ασφάλεια, την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλεια. Μιλήσαμε για την παρακολούθηση της γης, και τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Θα ήθελα να επανέλθω όμως και στην ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική. Δεν μπορούμε να προβάλλουμε ε, επιχειρήματα υπέρ μιας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, να μιλάμε για πρωταθλητές ευρωπαϊκής εμβέλειας, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι θα πρέπει να επηρεάσουμε την Κομισιόν, το Συμβούλιο και τους συναδέλφους της Επιτροπής Προϋπολογισμών για να γίνει αυτή η χρηματοδότηση είναι απαλήτως αναγκαία, αλλιώς δεν συμβαδίζουμε με αυτά που λέμε. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να δείξουμε αποφασιστικότητα και συνέπεια. Καρλ Σλίτερ. Άκουσα. Άκουσα τι είπε ο κύριος Πρόντι για τη χρησιμότητα όλων αυτών, αλλά νομίζω ότι δεν λειτουργήσε μια ιδέα περί συγχρηματοδότησης από κοινού με τη βιομηχανία και τώρα ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Γαλιλαίου και του GMS θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Και άρα τα κράτη-μέλη θα πληρώσουν για το αντίστοιχο στρατιωτικό σκέλος, έτσι, από τον προϋπολογισμό άμυνας. Εγώ προσωπικά αρνούμε να δώσω έστω και ένα σέντ για στρατιωτικούς σκόπους. Οποιαδήποτε διαστημική χρήση για στρατιωτικούς σκοπούς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς προϋπολογισμούς και όχι από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και σε καμία περίπτωση στα πλαίσια της διαστημικής μας πολιτικής θα πρέπει να προαγάγουμε μια στρατικοποίηση του διαστήματος. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκονζάλης τώρα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώνουμε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ήθελα μόνο να τονίσω ότι εφόσον ε, συζητούμε εδώ την ανακοίνωση 4 Απριλίου, θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει έλλειψη συνοχής ανάμεσα σε αυτήν και την προηγουμένη, δηλαδή στις 29ης Ιουνίου σχετικά με την ε, χρηματοδότηση των πολιτών προγραμμάτων. Στις 4 Απριλίου αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της την προτεραιότητα προγραμμάτων όπως το GMES και στις 29 Ιουνίου τονίζεται επίσης η σημασία αυτών των προγραμμάτων, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρέπει να χρηματοδοτηθούν διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται διάκριση ανάμεσα στο Γαλιλαίο, που, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαχειριστής και ιδιοκτήτη σε ποσοστό 100% και μην ξεχνούμε και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οπότε κάνουμε τη διάκριση με το GMES και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση για την χρηματοδότηση του. Δεν είναι ότι φάσκουμε και αντιφάσκουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις ή και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Υπάρχει μία πρόταση όπου εμπεριέχεται αυτή η ιδέα και προτείνεται η συνέχιση του GMES σε αυτό το χρηματοδοτικό πλαίσιο που ε, προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωση της 29 η Ιουνίου. Ε, κυρία Λεπάς, θα ήθελε ο εισηγητής ε, να προσθέσει κάτι. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στην Επιτροπή και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία αντίφαση, διότι θεωρούμε ότι αυτό το project είναι ένα κατά προτεραιότητα πρόγραμμα και δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Εφόσον πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα το οποίο προβάλλουμε κατά προτεραιότητα, θα, πρέπει, θα έπρεπε να είχε και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία είναι αύριο στις 6 για τις τροπολογίες, στις 25 θα ψηφίσουμε στο Στρασβούρου και ε, στις 23 Νοεμβρίου στη συνέχεια την έκθεση και τον Δεκέμβριο θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Θα περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ντανσέ για να μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση του, οργανισμού, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων. Σας περιμένουμε, κύριε Ντανσέ.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 Κυρίε και κύριοι, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Ευρωεπιτροπής Περιβάλλοντος, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εδώ για να σας ε, να κάνω τον ετήσιο απολογισμό του Οργανισμού για τις Χημικές Ουσίες του Ελσίνκη. Θα ήθελα να σχολιάσω όλους ιδιαίτερως τέσσερα στοιχεία, τα επιτεύγματα του 2010, κάποια στοιχεία κλειδί ε, για τις ε, μέχρι τούδε εμπειρίε μας, οι πολύ ενδιαφέρουσε προκλήσεις που μας περιμένουν και τέλος θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξή σας σε διάφορους τομείς. Μετά από αυτή την παρουσίαση θα έχουμε άπλετο χρόνο για να θέσετε όλα τα ερωτήματα που επιθυμείτε. Πρώτον, για τα επιτεύγματα, για τα περσινά μας επιτεύγματα. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι ενώπιόν σας και πάλι μετά από μια τόσο επιτυχημένη χρονιά για τον οργανισμό μας ε, και για τη φήμη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον ηγετικό ρόλο ε, στον τομέα των ασφαλέστερων χημικών ουσιών. Όταν συναντηθήκαμε πέρυσι, υπολείπονταν τρεις εβδομάδες πριν γίνει η πρώτη δοκιμή για την προθεσμία ταξινόμησης και καταχώρησης των επικίνδυνων χημικών ουσιών. Προχωρήσαμε λοιπόν στην κατα καταγραφή τους και θα ήθελα να σας Υπενθυμίσω ότι κάναμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και με επιτυχία ε, τηρήθηκε αυτή η προθεσμία ταξινόμησης και μετά από ένα μήνα τηρήθηκε και η προθεσμία σήμανσης για τις ε, χημικές αυτές ουσίες ε, τους τελευταίους μήνες του 2010 μπορεί κάποιος ε, αθώος παρατηρητής να θεωρούσε ότι καθόμασταν εκεί σαν πάπιες και επιπλέαμε πάνω σε ένα ποτάμι, σε ένα χήμαρο. Δεν ισχύει όμως αυτό διότι δεν μας βλέπατε, ήμασταν κάτω από το νερό και εργαζόμασταν άοκνα. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω ότι είμαστε ιδιαίτερη υπερήφανοι που ε, τηρήσαμε όλες αυτές τις ε, προθεσμίες. Ε, σχεδόν 25.000 φάκελοι κατατέθηκαν από χιλιάδες εταιρείε για τα πλέον κοινά και τις πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες στην Ευρώπη και υπήρξαν πάνω από 3 εκατομμύρια κοινοποιήσει για εξαιρετικά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Όπως σας είπα, ήδη πέρσι είχαμε την πεποίθηση ότι ήμασταν καλά προετοιμασμένοι και με το προσωπικό και το σύστημα πληροφορικής μας, αλλά φυσικά υπάρχουν πάντοτε αστάθμητοι παράγοντες, αλλά και πάλι στον οργανισμό μας ε, και σε συνεργασία με τους συναδέλφου ε, στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτή τη μέγιστη πρόκληση και έτσι καταστήσαμε ε, την Ευρώπη ασφαλέστερη. Ε, είμαι ευγνώμων ε, για όλους όσους συνεργάστηκαν, για όλους όσους μας συνεχάρισαν και είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας βοηθήσουν. Έχουμε διαδραματίσει λοιπόν το δικό μας ρόλο σε αυτό το σημαντικό επιχείρημα και αυτό θα ε, μας μείνει αξέχαστο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Επίσης, πέρα από ε, την Εκτελεστική Επιτροπή, έχουμε και το Διοικητικό μα Συμβουλίο που έχει ιδιαίτερη σημασία. Την περασμένη εβδομάδα λήφθησαν δύο στρατηγικέ αποφάσει. Πρώτον, το πρόγραμμα εργασία ε, για το επόμενο έτο ε, και θα δημοσιευθεί προσεχώ. Επίση, εγκρίθηκε η νέα πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων. Σίγουρα η Επιτροπή σα θα ενδιαφερθεί όλο ιδιαίτερο για αυτό το θέμα. Με ομοφωνία, λοιπόν, ελήφθησαν αυτέ οι αποφάσει και παρατάθηκε και η δική μου θητεία του εκτελεστικού διευθυντή Δηλαδή, ε, περατώνεται στα τέλη του 2012 κανονικά η θητεία μου και ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε την επιθυμία μου να υπηρετήσω για μια δεύτερη θητεία και τώρα ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να δρομολογηθεί δεν χρειάζεται να δρομολογηθεί νέα επιτροπή επιλογή και θα κάνουμε τα απαιτούμενα διαβήματα για να παραταθεί η θητεία μου. Α περάσω τώρα στο δεύτερο σημείο. Τι μάθαμε, ποια είναι τα διδάγματα. Ξέρετε ότι παράγουμε... Ε, έχουμε δημοσιεύσει δύο εκθέσεις ε, τον Ιούνιο του 2011 για την εμπειρία που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής και ο πρόεδρος μου ζήτησε να σχολιάσω αυτές τις εκθέσεις, οι οποίες είναι εκθέσεις στο άρθρο 117 για το ΡΙΤ και για το CLP και επίσης ε, τη χρήση εναλλακτικών χημικών ουσιών από πλευρά των επιχειρήσεων για το phasing out των δοκιμών στα ζώα. Ε, θα ε, ε, εκπονήσουμε πάντως και την πρώτη έκθεση για το Ρίτ. θα είναι η τελευταία χρησιμοποίησαμε αυτή την ευκαιρία για να εξετάσουμε ε, με διαφάνεια ε, και ειλικρίνεια την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει και να εντοπίσουμε τις ε, αδυναμίες και τα λάθη που κάναμε στο Ρίτσε. Επίσης, αποσκοπούμε στο να αγγίξουμε το ευρύτερο δυνατό κοινό και το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό των επιχειρήσεων που μπορούσαν να υποφεληθούν από τις εργασίες μας, γιατί οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι βασικοί δικαιούχοι του Ρίτσε και του και θα πρέπει να κατανοήσουν ότι σημειώνεται αυτή η πρόοδος ε, εξ ονόματός τους. Ε, σε 22 διαφορετικές γλώσσες ε, έχουμε εκλαϊκευμένες περιλήψεις των εργασιών μας, καθώς και σύντομα βίντεο στην ιστοσελίδα μας δείτε εδώ στον πίνακα τις εκθέσεις αυτές τις εκλαϊκευμένες, οποίες προανέφερα. Ε, και χάρη σε όλες αυτές τις κινήσεις όλο ε, ένα και περισσότεροι άνθρωποι ενημερώνονται για τα θετικά επιτέγματα στα πλαίσια του ΡΙΤΣ. Ε, το βασικό πόρισμα για το, την έκθεση του άρθρου 117 είναι πάρα πολύ απλό. Λειτουργεί το ΡΙΤΣ. Όταν δημιουργήθηκε το ΡΙΤΣ φοβόντουσαν κάποιοι ότι ήταν υπερβολικά φιλόδοξο, υπερβολικά σύνθετο, συνεπαγόταν μεγάλο βάρος διοικητικό και δημοσιονομικό για τις επιχειρήσεις, όμως το βασικό μήνυμα είναι ότι οι κανονισμοί, οι REACH και CLP λειτουργούν αισίως και ότι οι διάφοροι αρμόδιοι φορείς για αυτές τις εργασίες ανταποκρίνονται ε, όπως προβλέπει ο νόμος. Ε, σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της ε, νομοθεσίας μπορεί να αποδοθεί στην αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή βιομηχανία και άλλοι οικονομικοί φορείς, τα κράτη-μέλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οργανισμός μας. Όλες οι προθεσμίε από τον Ιούνιο το 2007 έχουν τηρηθεί ήδη και οι επιχειρήσει έχουν καταδείξει ότι δύναται να συνεργαστούν ε, και συχνά σε μεγάλου ομίλου εκατοντάδων επιχειρήσεων όπου ανταλλάσσουν δεδομένα και υπερβαίνουν οποιοδήποτε ενδιασμού είχαν για τη συνεργασία με τους ίδιους τους ανταγωνιστές τους. Ε, μόνο ε, κάποιε μεμονωμένε επιχειρήσει επιλέγουν από μόνε του να καταθέσουν τους φακέλους. Φυσικά όλα αυτά ε, δεν ήταν ε, απλά γιατί είναι μεγάλη η πρόκληση όταν ε, καλούμε να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε ένα νέο νομοθέτημα, αλλά γρήγορα αντλήσαμε τα διδάγματα και υπερβήκαμε τα εμπόδια. Ε, Παραδείγματο χάρη, συνειδητοποίησαμε ότι χρειάζονται συνεργατικές σχέσεις, σχέσει, επίση προδραστική επικοινωνία ανάμεσα στου συνυποβάλλοντε και διαφάνεια σχετικά με τι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα μέσα στο Ρίτσε και σε άλλα νομοθετήματα. Ε, και χρησιμοποιώντας έτσι ε, τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, και προγάγοντας τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίες καταφέρουμε να τηρήσουμε την πρώτη προθεσμία. Και παρόλα αυτά τα στοιχεία βασιζόμενοι στην εμπειρία και στη γνώση που είχαμε και τη σημασία αυτών των θεμάτων για τη σταθερότητα των επιχειρήσεων δεν προτείνουμε αναθεώρηση του κανονισμού Ρίτσε πριν εκπνεύσει η επόμενη προθεσμία φυσικά. Μικρή κλίμακα βελτιώσει ε, οφείλουμε να κάνουμε, αλλά θα έπρεπε η βασική νομοθετική σχέση να παραμείνουν αναλύωτοι αν θέλουμε να έχουμε ε, τις ε, μέγιστες δυνατότητες για την υποβολή φακέλων υψηλής ποιότητας μέχρι την εκπνοή της επόμενης προθεσμίας. Θεωρούμε ότι αυτό το έργο θα είναι ακόμη δυσχερέστερο για κάποιους νέους ε, για κάποιες νέες επιχειρήσεις ε, που έχουν στη διάθεσή τους ε, λιγότερα δεδομένα για νέες χημικές ουσίες. Θυμηθείτε επίσης ότι υπάρχουν και λιγότερο επικίνδυνες χημικές ουσίες οι οποίες παράγονται και τίθενται σε εμπορία σε μικρότερες ποσότητες. Και αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα. Στις Βρυξέλλες πριν από μία εβδομάδα έγινε μία διάσκεψη και καλέσαμε όλους τους ενδιαφερομένους να δράσουν ήδη τώρα και να αρχίσουν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την υποβολή των φακέλων για τις νέες χημικές ουσίες. Και πάλι για την εμπειρία μας ε, θα ήθελα να σχολιάσω τη δεύτερη έκθεση του άρθρου 117, δηλαδή σε ποιο βαθμό οι εταιρείε χρησιμοποιούν εναλλακτικέ χημικέ ουσίε για να αντικαταστήσουν τι δοκιμέ στα ζώα. Και εδώ είναι παρεμφερή τα δεδομένα, δηλαδή οι επιχειρήσει έχουν καταβάλει σοβαρότατε προσπάθειε για να χρησιμοποιήσουν τι διαθέσιμε εναλλακτικέ ε, μεθόδου ε, δοκιμών, ε, ούτω ώστε μόνο σε, σε ακραίε περιπτώσει να χρησιμοποιούνται αυτέ οι μέθοδοι δοκιμή σεζόν και προτείνονται 700, 700 διαφορετικές ε, δοκιμές ε, και έχουμε ξεκινήσει σχετικά μια δημόσια διαβούλευση ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει ε, καμία άλλη εναλλακτική μέθοδος. Έτσι θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις στις δοκιμές. Ξέρετε ότι οι πληροφορίες για την σε επιπτώσεις στους ανθρώπους και στο περιβάλλον είναι η κεντρική ιδέα, ο πυρήνας του Ρίτσε και πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον, αλλά και την ε, δυνατότητα, την ανάγκη να κάνουμε ε, δοκιμές, σε κάποια ε, ζώα όπως τα σπονδυλωτά παραδείγματος χάρη. Πάντως υπάρχουν ακόμη γκρίσες ζώνες. Ε, μία ανησυχία που είχαμε σε κάποιους ε, φακέλους ε, είναι η αιτιολόγηση που δίνεται από τις επιχειρήσεις. Συχνά η αιτιολόγηση για να βασιστεί μία επιχείρηση σε μία εναλλακτική μέθοδο δεν είναι τόσο κρατεά όσο θα θέλαμε. Εν τη αυτή περιπτώση αναπέμπουμε το φάκελο στην επιχείρηση και της ζητούμε να τεκμηριώσει πληρέστερα το φάκελό της. Φυσικά Μέτω χρειάζεται χρόνος ε, για να περατωθεί μια τέτοια διαδικασία, αλλά πάντως ε, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή αρχή και έτσι υπάρχει και καλύτερη ενημέρωση και μια καλύτερη εξασφάλιση για όλους μας σχετικά με την ασφάλεια στη χρήση των χημικών ουσιών στην καθημερινή μας ζωή. Τρίτο σημείο. Ποιε είναι οι εκπληκτικές προκλήσεις που μας περιμένουν στο μέλλον. Μετά την τήρηση των προθεσμιών για την ε, καταχώρηση και την κοινοποίηση μπορεί κάποιο να βρει δελεαστική, μια πιο παθητική στάση. Εν έχουμε άλλη προθεσμία πριν από δύο χρόνια μπορούμε να ε, ησυχάσουμε λίγο. Λυπάμαι, αλλά δεν αληθεύει αυτό. Θα σας πω ποιες είναι οι βασικές ε, προκλήσεις για το ECHA. Η πρώτη είναι να αξιολογήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους φακέλους ε, μπορούμε. Η αποτίμηση είναι σημαντική για το μέλλον του REACH. Σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που παράσχονται μέσα στις μεμονωμένους φακέλους. Επίσης όμως μας δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε ποιε ουσίες απαιτούν είναι περαιτέρω διαχείριση κινδύνου. Θέτει έναν ελάχιστο στόχο του 5% το ΡΙΤΣ, χωρί όμω να ορίζει χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν, ορίσαμε εμεί ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Το 2013 αποσκοπούμε στην αποτίμηση 5% των φακελών που έχουν κατατεθεί βάσει τη πρώτη προθεσμία καταχώρηση. Αν σα πω τώρα ε, ότι ένα φάκελο ε, για χημικέ ε, ουσίε επικίνδυνε και που τίθεται σε εμπορία σε μεγέθη, σε μεγάλο όγκο χρειάζονται 10.000 ε, περίπου διαφορετικέ επιστημονικές πληροφορίε. Καταλαβαίνετε πόση δουλειά συνεπάγεται αυτό. Χρειάζεται και πάλι εδώ μια ισορροπία ανάμεσα στους ενδεχόμενου κινδύνους ε, και τους επιλεκτικούς ελέγχους, ε, ούτω ώστε να μην έχει την εξασφάλιση καμία επιχείρηση ότι δεν πρόκειται να ελεγχθεί. Ε, επίσης, σε μία άλλη πρόκληση είναι ο εντοπισμός των ουσιών ε, ε, που μπορούν να προκαλέσουν ιδιαίτερη ανησυχία. Ξέρω ότι τα κάποια κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησαν αυτή την αδειοδοτική διαδικασία και ελπίζω ότι θα επισπευστεί. Αυτό επιθυμούμε και εμείς. Όλοι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, αλλά θα πρέπει να βλέπετε πιο γενικά τα πράγματα ο εντοπισμός ε, των ουσιών ιδιαίτερη ανησυχία είναι ένας μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, η πρώτη προθεσμία καταχώρησης ε, είχε ως αποτέλεσμα όλες οι καρκινογόνες ε, τοξικές ουσίες κατα, καταχωρήθηκαν και τώρα υπάρχει ένα μητρό που είναι διαθέσιμο για το κοινό στην ιστοσελίδα μας για πρώτη φορά. Και πάνω από τις μισές ουσίες ε, που είχαν ταξινομηθεί στο παρελθόν δεν είχαν καταχωρηθεί βάσει της πρώτης προθεσμίας και συνεχίζονταν ε, και εξακολουθούσαν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία να χρησιμοποιούν ευρύτατα αυτές τις ε, χημικές ουσίες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι τα πάντα ρίκη χρειαζόμαστε νέες πληροφορίες, νέα δεδομένα για την διαχείριση του κινδύνου για ε, τις ε, μεγάλες επιπτώσεις μπορούν να έχουν διάφορες χημικές ουσίες ε, όπως αυτές που επηρεάζουν το ενδοκρινικό μας σύστημα. Μία άλλη πρόκληση είναι ε, αυτή της ενημέρωσης. Ε, μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου η ε, ECHA είχε δημοσιεύσει πληροφορίες σχεδόν για όλες τις ουσίες που είχαν καταχωρηθεί βάσει της προθεσμίας του 2010. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε αυτό τον πακτολό πληροφοριών που έχουμε στην ιστοσελίδα μας και να βρούμε τη βέλεστη δυνατή ισορροπή οποία ανάμεσα στη δημοσίευση στο μέτρο του δυνατού και την ε, προστασία τη ε, βιομηχανία. Δηλαδή, οι τεχνικέ και επιστημονικέ αυτέ πληροφορίε, ναι, μεν πρέπει να είναι διαθέσιμε για το ευρύ κοινό, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τι δυσκολίε ε, που ανέχει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να προ... επιτύχουμε μια καλύτερη κατανόηση από πλευρά όλων των ενδιαφερομένων. Η πέμπτη και τελευταία πρόκληση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ έχει ιδιαίτερη σημασία για σας. Ε, δηλαδή, οι ευθύνες ε, που φέρουμε βάση ε, των επικείμενων κανονισμών ε, για τα βιοκτώνα ε, και για τις χημικές ουσίες για τις οποίες χρειάζεται πρώτερη έγκριση. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτούς τους κανονισμούς και φυσικά θα επιταχύνουμε τις δραστηριότητες μας μετά την έγκριση του κανονισμού όταν θα έχουμε και τους απαιτούμενου πόρους. Παρακολουθούμε εκ του και στην νομοθετική διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νιώθουμε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για την Επιτροπή Περιβάλλοντος διότι στην πρώτη πρόσφατη ανταλλαγή απόψεων που έγινε για την, το σχέδιο Έκθεση τη κυρία Κλά για το ECHA μας προσκαλέσατε να παραστούμε. Και περιμένουμε φυσικά και με αδειμονία τα αποτελέσματα της δεύτερης ανάγνωσης για τον κανονισμό για τα βιοκτώνα σήμερα. Ε, επίσης ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για το 2010. Μιλήσαμε για τις εμπειρίες και τώρα φτάνω στο τελευταίο σημείο. Σε ποιους τομείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια και την υποστήριξή σας. Ε, πρώτον, θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε την επιρροή που έχετε σε εθνικό επίπεδο. Το REACH βασίζεται στην δυνατή στενή συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κέριος ο ρόλος των κρατών μελών, όχι ως προς την υποστήριξη που προσφέρουν στη βιομηχανία και την ενίσχυση νομοθετικής διαδικασίας, αλλά και ω προ ε, την διαδικασία λήψη επιστημονικών αποφάσεων. Είναι κρίσιμη η κατάσταση, υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί που όλοι ξέρουμε και χωρί ε, του απαιτούμενου πόρου σε εθνικό επίπεδο ε, ενδέχεται να θέσουμε σε κίνδυνο την επιτυχία του ΡΙΤΣ. διότι το επίπεδο της τέχνογνωσίας ως προς τι χημικέ ουσίες σε επίπεδο κρατών μελών είναι μια πηγή ανησυχία. για μα. Χρησιμοποιήστε λοιπόν την επιρροή που έχετε σε εθνικό επίπεδο για να συνεχίσει να ε, συνιστά προτεραιότητα το REACH. Δεύτερον, ε, θα ήθελα να μας βοηθήσετε ε, ως προς την ενημέρωση των επιχειρήσεων στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες για την ευθύνη που φέρουν. Κυρίως αναφέρομαι στις μικρές επιχειρήσεις. Εάν ε, χρειάζεστε κάποια βοήθεια να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Ε, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την τήρηση της επόμενης προθεσμίας ε, το 2013 γιατί τότε θα καταχωρηθούν για πρώτη φορά πολλές νέες επιχειρήσεις. Πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε η εκστρατεία ενημέρωσης του ECHA και τυπλοφορείται REACH 2013 δράστε τώρα και αυτό πρέπει να κάνουν ακριβώς οι επιχειρήσεις. Βοηθήστε μας να ενημερώσουμε τις επιχειρήσεις. Λοιπόν, τέλος, οι μας, όπως ξέρετε, ε, χρεώνουμε τις υπηρεσίες μας ε, στην βιομηχανία Ζητούμε τέλεια από τις επιχειρήσεις και δεν χρειαζόμαστε υποστήριξη από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αποθεματικά στην τράπεζα και θα μπορέσουμε να καλύψουμε το κόστος ε, των εργασιών μας για τα ερχόμενα χρόνια. Όμως το 2014 θα έχουν εξαντληθεί αυτά τα αποθέματα και για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε θα ε, χρειαστούμε για τον επόμενο χρηματοπιστωτικό κύκλο χρηματοδοτική υποστήριξη. Αυτό δεν είναι κάτι ε, καινούριο ή απρόβλεπτο, αλλά αντιστοιχεί στον ε, ε, οικονομικό σχεδιασμό του ΡΙΤΣ ε, που επιλέξατε εσείς και το Συμβούλιο όταν εγκρίνατε το σχετικό κανονισμό το 2016. Οπότε απευθύνω θερμή έκκληση προς εσάς να το έχετε κατά νου όταν εξετάσετε τα κονδύλια για την περίοδο 2014-2020. Είναι το πλέον σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για τις χημικές ουσίες στον κόσμο το ΡΙΤΣ και θα ήθελαμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας, να υποστηρίξουμε την κυρία Χάουκ που πρότεινε 10 νέες γραμμές για το ECHA για του χρόνου. Θα, θα χρηματοδοτούνται αυτά βεβαίως από, οι 10 αυτές νέες θέσεις θα χρηματοδοτούνται από τα τέλη και όχι από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ελπίζω στις τελικές συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2010 να υποστηρίξει αυτή τη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και στις επόμενες διαπραγματεύσεις για την περίοδο μέχρι το 2020. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δώσατε ε, να υποβάλω αυτή την αναφορά για τι δραστηριότητε ε, του οργανισμού μας ε, και περιμένω με αγωνία τα σχόλιά σας. σας... Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Πολλές ερωτήσεις ασφαλώ θα προξενήσουν οι παρατηρήσει σα από πλευρά των συναδέλφων. Μπορούμε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης, τη προόδου, του τι δρόμου που έχουμε είσουμε ακόμα. Το λόγο. Α λάβει πρώτη η κυρία Χάση. Ως εκπρόσωπο μα στην υπηρεσία σας. Πρώτη παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Λάνσετ. Να μας δώσετε στοιχεία για τη δουλειά της υπηρεσίας σας. Όπως είπατε κι εσείς, έχει τεράστιο έργο και ιδιαίτερα στη διερεύνηση τη κλιματική Αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα ως προς την εφαρμογή του REACH. Αν και θα περιοριστώ σε ένα μόνο αυτή τη στιγμή. Ποιότητα των στοιχείων φακέλων, δηλαδή προς καταχώρηση, που διαθέτει η βιομηχανία. Ε, είπατε εσείς ότι ελπίζετε πως θα είναι καλύτερος, καλύτερη ποιότητα στο μέλλον. Στην πρώτη πενταετία αναφέρεται ότι μεγάλο αριθμός φακέλων προς καταχώρηση επαληθεύονται και υποδεικνύεται ότι δεν τηρούν πλήρως τι προδιαγραφέ ή δεν υπάρχουν επαρκέ πληροφορίε. είτε δεν υπάρχουν επαρκε πληροφορίες, είτε η ποιότητα των παρχομένων πληροφοριών είναι ανεπαρκής. Για να στεφθεί όμω με επιτυχία το REACH, να λειτουργήσει πραγματικά, το πιο σημαντικό πιστεύω και η θεμελία αλήθως είναι να υπάρχουν ακριβή στοιχεία. ακριβή στοιχεία δεν είναι ευθύνη της βιομηχανία να προσφέρει. Ξέρουμε ότι στην αρχή της προσπάθειας μόνο τα μισά από τα απαιτούμενα έγγραφα παρουσίαζαν πρόβλημα. Ερωτώ λοιπόν, η υπηρεσία χημικών ουσιών τι κάνει Πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα των ανεπαρκώς στοιχειοθετημένων ε, φακέλων, πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό, ώστε να ξέρει και όποιος χρήστη ότι μπορεί να εμπιστεύεται τα στοιχεία που συμβουλεύεται. Και επίσης μιλάτε για ένα 5% των φακέλων. Ερωτώ λοιπόν σε ποιο βαθμό η ανεπάρκεια αυτή, οι ατέλειες αυτές τους υποβλημένους ε, φακέλους προξενεί και ε, καθυστερήσεις με την έννοια της ε, τελικά, του τελικά ελληπούς ελέγχου των φακέλων. Κυρία Γκροστάτε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας παρουσιάσετε τον απολογισμό σας, αλλά και τις προοπτικές για το μέλλον ενός κανονισμού που μας είχε απασχολήσει για πολλά χρόνια. Θα ήθελα απλώς να σας επισημάνω, μια και μας παρουσιάσετε με τόσο θετικό τρόπο τον απολογισμό σας, και πολύ καλά κάνατε, κανείς δεν αμφισβητεί αυτή τη χρησιμότητα αυτού του κανονισμού. Απλώς πιστεύω ότι αυτά τα οποία ε, βλέπουμε συχνά δεν είναι τόσο θετικά. Και δεν μιλάω για τις μεγάλες επιχειρήσεις που σε τελευταία ανάλυση έχουν κάθε τρόπο να χειριστούν το θέμα αυτό. Όχι, μιλάω για τις ε, πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα του κανονισμού REACH. Θα ήθελα λοιπόν γιατί πω ένα συγκεκριμένο ερώτημα που αφορά και την ε, δική μου ε, εκλογική περιφέρεια. Ε, αυτούς που ασχολούνται με την ε, παραγωγή και απόσταξη αρωμάτων και ιδιαίτερα όσους έχουν να κάνουν με εθέρια έλαια. Και ε, οι επιπτώσεις του ρίτς σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το τομέα της παραγωγής, γιατί είναι μεν αφορά ουσιαστικά τις χημικές ουσίες, αλλά εφαρμόζεται από την άλλη στην πράξη στα φυσικά, στα εθέρια έλαια, πράγματα, πράγματα τα οποία είναι ως εκ της φύσεως τους φυσικά προϊόντα, Ωστόσο, πρέπει να καταχωρήσει ε, με βάση το REACH με κόστος 150.000 περίπου ευρώ ανά ουσία και είναι τόσο πολύ μεγάλο η αποτρεπτική δύναμη αυτού του κανονισμού και της οικονομικής επιβάρυνσης που επιβάλλει που μπορεί να χαθούν ορισμένες επιχειρήσεις μόνο και μόνο γιατί δεν είναι σε θέση να καταχωρήσουν για κάθε εθέριο έλαιο που χρησιμοποιούν διαφορετικό φάκελο. Για δε την τοξικότητα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαδικασία αξιολόγησης. Είναι ελάχιστη η κίνδυνη, ούτως ή άλλως όπως σας είπα πρόκειται για φυσικές ουσίες, ουσίες που αντλεί κανείς από την ίδια την φύση. Οι ρηπαντικές τους ιδιότητες είναι πολύ περιορισμένες. Οι δε υποχρεωτικές αναφορές που θα πρέπει να υπάρχουν στην ε, σήμανση του προϊόντος, στην ετικέτα δηλαδή δυνάμει του κανονισμού REACH, προβλέπουν φερρυπίν για τα εθέρια έρλια, για το εθέριο έρλιο της Λεβάντας που είναι γνωστό <laughs> από την αρχαιότητα χρησιμοποιείται ως τις μέρες μας. Καταγράφεται λοιπόν, καταχωρίζεται μάλλον στην κατηγορία πολύ τοξικό για το υδάτινο περιβάλλον. Το εθέριο έλαιο της Λεβάντας. Ναι, μπορεί για το, εθέριο, για το, για το θαλάσσιο περιβάλλον μία σταγόνα Λεβάντας να μπορεί να οδηγήσετε σε θάνατο ένα ψάρι σε ολόκληρο τον ωκεανό ή ένα δέντρο σε ολόκληρη τη γη, αλλά μήπως είναι υπερβολικέ οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού Ρίτζ για κάτι τόσο απλό και τόσο μηδαμινό. Γιατί μιλάμε για μια μικροσταγόνα. Και επίση θέλω να σημάνω ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα σημαντικό και οικονομικό για όλη μου την, ε, για όλη μου την εκλογική περιφέρεια που έχει στη νοτιοδυτική Γαλλία την, ε, τον κύριο όγκο της παραγωγής Λεβάντας και γενικά θερίων ελαίων και που η ε, αγωνία θέλει να εισακουστεί η φωνή της, θέλει να γίνουν κατανοητές οι ανησυχίες και οι αγωνίες της. Και δεν την απάντηση σας παρακαλώ. Ευχαριστώ Χριστίνης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να αναφερθώ και στην παρατήρηση της κυρίας Χάση για το 50% των φακέλων που αναφέρθηκε. Ε, όταν έχετε τόσες προϋποθέσεις επαλήθευσης, ε, στην επαλήθευση κάθε, των φακέλων όταν υπάρχουν τόσες προϋποθέσεις, προφανώς θα, θα βρείτε κάπου σφάλματα. Είναι δύσκολο να ξεσφαλιστεί κάποιος φάκελος αλάνθαστος, άμεμπτος. Άρα τι έχετε δαχθεί από την μέχρι τώρα εφαρμογή του συστήματος. Επίσης για την ε, αλυσίδα παραγωγής και την κρίση των ουσιών. Τι βλέπετε. Εν γέννη θα ήθελα να σημειώσω ότι έρχεται στην Επιτροπή μας δίνεται μια πολύ θετική εικόνα. Τόσο θετική θα έλεγα που εγώ τίνω στον κινησμό ε, με την μόνη παρένθεση ότι δεν μου έχει γράψει κανείς από τη χημική βιομηχανία της περιοχής μου στην ε, Αγγλία Πράγμα το οποίο με δύο τρόπου εξηγείται. Ή είναι ευχαριστημένοι από την εφαρμογή του Rich ή έχουν χάσει την διεύθυνσή μου την ηλεκτρονική και δεν μπορούν να μου στείλουν email. Εν πάση περιπτώσει, παρά τα σχόλια της Φωνσουάς Κροστέτ ότι δεν αμφισβητεί κανείς τους λόγους για τους οποίους έχει επιβληθεί, έχει θεσπιστεί αυτός ο κανονισμός REACH, καθώς εγώ προέρχομαι από χώρα πολύ επιφυλακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη διάσκεψη στην οποία αφισβητείται κάθε τύπου κανονισμός και νομοθεσία ω ε, προ ως προς την χρησιμότητά τους. Ερωτώ λοιπόν, ε, ναι, πολύ καλή δουλειά που κάνετε, πολύ καλό το προϊόν της εργασίας σας, αλλά δεν νομίζετε κι εσείς ότι το REACH επιβάλλει υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό οδηγεί σε δυσμενέστερη τοποθέτηση ως προς την ανταγωνιστική μας θέση. Και υπερβολικά σημαντικές πιέσεις εις βάρος των επιχειρήσεών μας που δεν έχουν σε τελευταία το όργανο μικρομεσαίων, που δεν έχουν σε τελευταία ανάλυση και το, ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε την τεχνικό, υλικοτεχνική υποδομή για να απαντήσουν ε, σε αυτά. Είναι λοιπόν, θα έλεγα, η ερώτησή μου κάτι σαν τη θέση του συνεγόρου του διαβόλου, γιατί κατά τα άλλα εγώ συμπαθώ ιδιαίτερα το Ρίτς, αλλά έπρεπε να ρωτήσω. Dans l'autre sens. Madame vous voulez... Κυρία Κλάς, εσείς έχετε τίποτα να πείτε. σκένε, λόγο ο κύριος πρώτος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Τάνσερ, που βρίσκεται εδώ μαζί μας και να υπογραμμίσω τη σημασία του Ρίτς, διότι πράγματι είναι ένα στοιχείο αναφοράς για την ασφάλεια στα εργαστήρια αλλά και στο περιβάλλον γενικότερο, γενικότερα. Θα ήθελα να παρέμβω για να ζητήσω βοήθεια και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό αυτό. Εγώ είμαι μέλος της ΣΤΟΑ που αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία, την αξιολόγησή τους και θα ήθελα να του πω ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένες έννοιες έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται σωστά στο στη νομοθετική γλώσσα. Ιδιαίτερα όταν αξιολογούμε τους κινδύνους, όταν κοινοποιούμε τους κινδύνους, ζητώντας από, όλες, από όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς να συνεργαστούν, διότι έχουμε να κάνουμε με μία άμεση ανάγκη να είμαστε πιο ευκρινείς είτε στη λειτουργία του κάθε οργανισμού, είτε ως προς την ανάγκη να έχουμε κοινή θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, αυτό το συμπλήρωμα της αξιολόγησης του κινδύνου είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει δηλαδή να βαστούμε στην αρχή της ε, πρόληψης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τελειοποιηθεί γιατί θα μπορούσε να μας ε, βοηθήσει περαιτέρω. Θα ήθελα να προανακοινώσω αυτό το αίτημα, το οποίο θα γίνει προς όλους τους οργανισμούς για αυτή την κοινή προσπάθεια, έτσι ώστε να ορίσουμε μια ενιολογική βάση και να χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την επιστημονική μας κοινότητα. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Ελπίζω να μην με... Ε, ελπίζω να με είδατε, ελπίζω να με παραβλέψατε. Εν πάση ευχαριστώ πολύ και για τις πολύ αισιόδοξε και γεμάτε αυτοπεποίθηση παρατηρήσεις. Καλό κάνει να ακούμε ότι δουλεύει καλά το REACH και ότι έχει πάρει το ρυθμό του, λειτουργεί καλά Έχουμε το θέμα των βιοκτώνων και θα ήθελα να ρωτήσω εγώ ως αρμόδια εισηγήτρια τι είδους συνεργατικές σχέσεις μπορούμε να έχουμε στο θέμα των βιοκτώνων. Αύριο θα μας απασχολήσει η ψηφοφορία της σχετικής έκθεσης. Και επίσης καλό θα ήταν να μας πείτε πώς ενδεχομένως μπορούν να συνδεθούν τα θέματα αυτά μεταξύ τους, δεδομένου ότι όταν έχουμε αποδεθεί στην ίδια προσπάθεια και έχουμε κοινό υλικό να επεξεργαστούμε, ε, καλό θα είναι να έχουμε συνεργατικές ε, σχέσεις. Θα ήταν καλό δηλαδή να τα βλέπουμε όλα αυτά μαζί. Επίσης θα ήταν καλό να κοιτάξουμε και το θέμα του κόστους. Τη αιτήσια τέλη, την αιτήσια επιβάρυνση, η πρόσθετη επιβάρυνση δεχομένω. Και βεβαίω ε, αυτό το οποίο ανέφερε η κυρία Γκροστέτ είναι πολύ σημαντικό γιατί μερικέ φορέ δεν είναι δυνατόν να προεξοφλούμε ότι κάθε φυσικό προϊόν, κάθε προϊόν της φύσης είναι ακίνδυνο, δεν χρειάζεται καταχώρηση. Άρα κάποιο τύπου καταχώρηση θα χρειάζεται φαντάζομαι ακόμη και για τα φυσικά προϊόντα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε μια διάκριση, να υπάρχει μια διαφορετική, ένας διαφορετικός χειρισμός ακόμη και προς το θέμα των τελών, της ε, συμμετοχής δηλαδή για τις φυσικές αυτές ουσίες. Το ίδιο ισχύει ασφαλώ και για ουσίε, οι οποίε δυνάμει άλλων κανονισμών ή οδηγιών ε, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται. Ε, Φερρυπίν, ε, ουσίες ε, όπως το διοξίδιο του θείου που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την κονσερβοποίηση ως πρόσθετο στα τρόφιμα. Εάν είναι λοιπόν ως πρόσθετο στα τρόφιμα επιτρέπεται η χρήση του, εάν όμως χρησιμοποιείται ως βιοκτόνο, τότε χρειάζεται επιπλέον αδειοδότηση με πολύ υψηλό κόστος, μέχρι και 150.000, από 150 μάλλον μέχρι 500.000 ευρώ το κόστος για τη χρήση, πράγμα το οποίο βέβαια οδηγεί σε πολύ ασαφείς ε, συνθήκες ε, νομοθετικές για την κάθε ουσία, πράγμα το οποίο καθόταν καλό να συζητήσουμε και να αποφύγουμε βεβαίως ε, τον πολλαπλασιασμό των νομοθεσιών και των σχετικών επιβαρύνσεων. Δεν ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα έχουμε να κάνουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για τον κύριο Chris Davis επίσης ήθελα να πω ότι σε μεγάλο βαθμό φταίμε και εμείς, γιατί και τα κράτη-μέλη πολλές φορές, δηλαδή οι διοικοί των κρατών μελών πολλές φορές περιπλέκουν τα πράγματα και ζητούν όλο και πιο πολλές πληροφορίες. Ε, όπως σε παραδείγμα, οι ενδοκρινικές ε, δομές είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει Τώρα Θέλουμε να έχουμε όλο και πιο πολλά στοιχεία και να ε, ενημερωνόμαστε όλο και περισσότερο. Πολλά είναι τα ερωτηματικά λοιπόν στον τομέα αυτών. Και καλό θα ήταν να ε, μπορούμε να προσμετρήσουμε την ε, αξία αυτών των ουσιών. Και ελπίζω ότι στο μέλλον, όταν θα έχουμε και τις νέες μεγάλες προκλήσεις, το Ρίτσι θα είναι πάλι σε θέση να δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ, Σλίτσας. Yeah. Hi and welcome. Γεια σας και να σας καλωσορίσω κι εγώ. Έχω έχω τρία ερωτήματα. Εγώ σας είχα ρωτήσει πόσα, ε, ε, πόσους φακέλους έχετε εγγεγραμμένους και εσείς μου είπατε ότι είναι τρεις. Ως προς το, την ποιότητα και τις παρατηρήσεις και όταν βλέπετε ότι η στοιχεία δεν λείπουν αλλά δεν είναι σωστά, τι κάνετε. Επίσης αποστήλατε αρκετές επιστολές τέτοιου είδους και είδατε τα προβλήματα ή την ποιότητα των φακέλων. Ίσως θα πρέπει να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα και να ζητήσουμε με τη συνεργασία των κρατών μελών να δούμε ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι ελληματικές στα στοιχεία. Δηλαδή λένε μόνο το 5% θα εγκριθεί, άρα δεν χρειάζεται να δώσουμε όλα τα στοιχεία όλων των φακέλων. Είδατε είδατε να υπάρξουν κυρώσεις ή χρηματικές ποινές κατά επιχειρήσεων που δεν συμμορφώθηκαν. Και ίσως και αυτό θα ήταν ένα μέτρο συμμόρφωσης. Σε σχέση με τον κατάλογο υποψηφίων, πώς θα φτάσετε στο στόχο των 136 και γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος για την Επιτροπή τη στιγμή που θέλετε να κινηθείτε στο παράρτημα 15 τη στιγμή που μία επιχείρηση φαρμάκων υποβάλλει ε, μία αίτηση, συνήθως η Κομισιόν αποφασίζει αμέσως. Εσείς πώς κινείτε την διαδικασία αδειοδότησης ή απαγόρευσης, γιατί είναι τόσο χρονοβόρος η διαδικασία. Δηλαδή μετά από την κρίση σας θα έπρεπε να είναι πολύ γρήγορη απόφαση. Η Άννα Ρόσπαχ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις μέχρι τώρα προς τον κύριο Ντάνσετ. Δεν έχω να προσθέσω πολλά, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τη στιγμή που το REACH δεν εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη, τι κάνετε εσείς για να γίνει η σωστή εφαρμογή του κανονισμού REACH στα 27 κράτη-μέλη, γιατί τότε αν δεν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσα προσκόμματα υπάρχουν σε επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Έχετε κάποια γνώμη γιατί εμείς είμαστε πιο αυστηροί ε, εμείς σε σχέση με την Κίνα, τη ΣΥΠΑ και την Ιαπωνία. Merci, Η Σοφία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Ντάνσετ για την σαφήνεια της εισήγησής σας. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους και ιδιαίτερα με τη Φρανσουάς Γκροστέτ γιατί πράγματι θα πρέπει να εργαστούμε επί της ουσίας ως προς το θέμα του κανονισμού, του ρυθμιστικού πλησίου σε σχέση με την χημική ουσία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τα πάντα. Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση. Όμως έχουμε ΜΜΕ που δεν έχουν τις ε, κατάλληλες, ε, την κατάλληλη υποδομή για να μπορέσουν να ε, δεχτούν αυτές τις ρυθμίσεις πέρα από τις ρυθμίσεις που, που ισχύουν για το περιβάλλον. Πρόκειται και ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη φορολογία και οδηγίες που μεταφέρονται στα κράτη-μέλη αλλά οι μικρές επιχειρήσεις δεν ξέρουν πώς ε, μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ε, αλληλοστρωμάτωση των ε, ρυθμίσεων. Θα πρέπει λοιπόν στον τομέα της ρύθμισης να μην ασχολούμαστε, να μην, να μην έχουν αυτές οι ρυθμίσεις πολλαπλαστή πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, έτσι ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μην πλήττονται ως προς την ανταγωνιστικότητά τους, διότι αυτές οι ρυθμίσεις πολλές φορές είναι επαχθείς, επαχθέστερες σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σνίμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι πολύ καλά την εποχή που φτιάχναμε το Rich. Είναι καλό που βλέπω και τον κύριο Σακόνη εδώ. Ήταν ε, στιγμές ε, ανατρεπτικές. Ε, λεγότανε ότι θα ανατραπεί το πεδίο της χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Και όμως δεν υπάρχουν προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Επανλήθευσε και ο κύριος Κρις Ντέιβις που λέει ότι δεν λαμβάνει μηνύματα παραπώνων από την χημική βιομηχανία. Το είδα και εγώ μέσω των συνεργατών μου. Φαίνεται ότι πάει καλά το ε, REACH. Μπορούμε να είμαστε εν γέννη περήφανοι παρά τα κάποια μικροπροβλήματα που επισημαίνουν κάποιοι συνάδελφοι και μπορείτε να είστε και εσείς υπερηφάνος για τη δουλειά που κάνετε στην υπηρεσία χημικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ζήτημα όμως παραμένει εκρεμές είναι αυτό της γλώσσας. Σας το είχα θίξει και την προηγούμενη φορά. Ξέρω ότι εδώ μεταξύ έχουν εκείνη πολλές μεταφράσεις, αλλά πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ήθελαν να περισσότερη ε, δυνατότητα πρόσβασης ε, στις οδηγίες, στις γλώσσες τους. Για τόση επί Κρίστα Κλάς το καθεστώς των τελών της συμμετοχής είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, σχεδιαστεί κατά τρόπο πιο διαφανή πιστεύω, να λειτουργήσει κατά τρόπο πιο διαφανή γιατί είπατε και εσείς ότι τα τέλη είναι αυτά που χρηματοδοτούν τη λειτουργία σας μας είπατε με, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερος ότι έχετε και αρκετά χρήματα, πολύ καλά ε, βλέπουμε Ωστόσο ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και η διαφάνεια για τον ε, τρόπο με τον οποίο ε, χρηματοδοτήσετε. Δεν είσαστε τράπεζα στη τελευταία ανάλυση, δεν πρόκειται να κάνετε τις επενδύσεις μακροπρόθεσμα για να έχετε απόδοση. Ε, θα ήταν καλό λοιπόν να συζητήσουμε λίγο πιο ξεκάθαρα το θέμα των τελών, ιδιαίτερα προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κάτι για τον κύριο Εφηντή. Ίσως θα ήταν καλό να συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο, ή μάλλον το επίπεδο στο οποίο γίνεται η δουλειά, υψηλό επίπεδο ε, προστασίας καταναλωτή, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος είναι δουλειά δική σας μαζί με τις κυβερνητικές οργανώσεις δηλαδή μπορείτε και πρέπει να κάνετε αυτή την προσπάθεια και άπαξ και έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα του REACH, νομίζω ότι μπορείτε και στο επικοινωνιακό πεδίο να δραστηριοποιηθείτε περισσότερο για να κατανοήσει και ο πολίτη πολίτης ότι δεν κινδυνεύει κάθε μέρα από δηλητηρίαση επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά χημικά και επικίνδυνες ουσίες. Σε πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορείτε και επικοινωνιακά να δώσετε μια θετική ε, νότα στη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ και πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ντάνσετ που θα απαντήσει στα ερωτήματα που ακούστηκαν. Θα παρακάσω τον κύριο Γκουίτο Σακόνη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκπρόσωπος ε, του, στο Διοικητικό Συμβουλίο της Υπηρεσίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και όλους τους ε, συναδέλφους που ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα άλλη μια φορά. Θα είμαι πολύ σύντομος διότι ο εκτελεστικός σύμβουλος, ο κύριος Ντάνσετ, ε, μας έδωσε πολλές λεπτομέρειες. Ε, ως πρώην συνάδελφος θα ήθελα να πω ότι αν κάτι δεν πάει καλά με τον κανονισμό, φταίει ο νομοθέτης και καταρχήν εγώ γιατί εγώ πρωτοσυνέταξα αυτό το κανονισμό. Όμως εδώ συζητάμε πώς εφαρμόζεται ο κανονισμός αυτός σε σχέση με αυτό το μέσο το οποίο δεν υπήρχε πριν και τώρα, μάλλον εδώ και λίγο καιρό έχει συσταθεί, δηλαδή ε, μιλάω για τον ορισμό του Ελσίνκη. Δεν θέλω να ε, υπερβάλλω και να αρχίσω τις ε, θριαμβολογίες. Πιστεύω όμως ότι τα πράγματα πάνε καλά, καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το REACH ε, αφορά 45 οδηγίες που συγχωνεύτηκαν πριν και δεν λειτουργήσαν εδώ και 25 χρόνια. Γι' αυτό Μιλήσαμε για κάτι μεταξύ 300 και 400 ουσιών και με βάση τις πρώτες εγγραφές, η πρώτη εγγραφή έληξε λίγο καιρό πριν σε σχέση με ε, αυτά τα στοιχεία ως προς, και ως προς την ενημέρωσή τους. Τώρα βλέπουμε ότι είναι χιλιάδες 5.000 τουλάχιστον οι ουσίες που έχουν καταγραφεί. Άρα έχουμε μία τεράστια βάση δεδομένων όπου όλες αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται και κοινοποιούνται κιόλας. Γύρω στη, μιλάω για γύρω στις 3.000 Πρόκειται για ουσίες ε, στις οποίες μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση. Νομίζω λοιπόν ότι το σύστημα, οι προειδοποιήσεις που αποστέλει ο οργανισμός της επιχειρήσεις ως προς που δεν είναι πιστικά, όλα αυτά οδηγούν σε μέρους ανακτήσεις από αυτό το φαινόμενο. Η επόμενη προθεσμία του 2013 αφορά ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρήσεων με πολύ, μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερες, ε, μεγαλύτερα ποσοστά. Γιατί εμείς τι κάναμε, ιεραρχήσαμε το σύστημα έτσι ώστε όσο πιο μεγάλο να είναι το ΝΑΣ τόσο μεγαλύτερο να είναι και το ενδιαφέρον μας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις για να μην έχουν αυτό το γραφειοκρατικό άχθος. Και αυτό το θέμα αρχικά είχε δημιουργήσει πρόβλημα στην επιχείρηση, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διάφορες συμπράξεις, κοινοπραξίες και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να πω ότι ότι βεβαίως εγώ έχω ε, περιορισμένη ευθύνη πλέον, αλλά θα ήθελα να πω στον κύριο Ντάνσεστ ότι όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί δεν σταμάτησε ποτέ αυτή η διαδικασία. Θα ήταν απαράδεκτο να μην ε, ε, προβάλλουμε τροποποιήσεις, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να είναι πρόορες σε σχέση με την ε, πείρα μας. Γιατί υπάρχουν και άλλες μεταγενέστερες φάσεις μετά την αδειοδότηση. Έχουμε και την αξιολόγηση σε σχέση με την τοξικότητα των ουσιών και εδώ τα κράτη-μέλη φέρουν μεγάλη ευθύνη θα πρέπει να αναλάβουν δηλαδή την αξιολόγηση αυτών των ουσιών. Νομίζω ότι θα ήταν μου να αναπτύξουμε, να επιταχύνουμε αυτή τη μηχανή χωρίς όμως να προδικάσουμε την έκφαση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έξι χρόνια πριν όλα αυτά ήταν αδιανόητα γιατί είχε γίνει λόγος ε, ότι θα καταδικάσουμε τη χημική βιομηχανία. Αυτό λεγόταν, αυτό το λέω εν είδη αστείου βεβαίως. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα που θέλουν να προβούν ε, σε αυτή τη ρύθμιση. Δεν είναι αντίγραφο του δικού μας REACH, αλλά εν πάση χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν σαν βάση το δικό μας σύστημα REACH για να εκπονήσουν ένα δικό τους σύστημα. Γιατί το REACH βοήθησε και στην ανταγωνιστικότητα των ε, ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Άκρος ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Ίσως ο κύριος Βίλμοτ θα ήθελε το λόγο και μετά ο κύριος Άνσεντ από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Η Κομισιόν έχει το λόγο, όπως θέλετε, με τη σειρά που επιθυμείτε εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε ως προς ένα σημείο υπήρξε ένα ερώτημα προς τον κύριο Ντάνσετ που αφορούσε περισσότερο κομισιόν. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να περάσουν αυτές οι ουσίες στο παράρτημα 14 και γιατί η Επιτροπή δεν ε, ε, λειτουργεί πιο γρήγορα. Ε, λαμβάνουμε τις προτάσεις από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και μετά θα πρέπει να ε, κάνουμε εμείς τις ρυθμίσεις με βάση ένα κανονισμό. Γίνεται μία ε, συζήτηση μέσα στην Επιτροπή και επιλύουμε τα επιμέρους θέματα και κοινοποιούμε το θέμα στο, στον ΠΟΕ γιατί υπάρχουν ενδιάμεσα στάδια μετά ψηφίζεται από την Επιτροπή ΡΙΤΣ και χρειάζεται να παρέλθουν τρεις εβδομάδες, μετά αποστέλλεται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για εξέταση που μπορεί να επεκταθεί μέχρι τους τρεις μήνες. Μετά εγκρίνεται ο κανονισμός της Επιτροπής και χρειάζεται μία ή δύο εβδομάδες έτσι ώστε να φτάσουμε στην απόφαση. Άρα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ε, βήματα τα οποία είναι απαραίτητα και γι' αυτό πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος για να ενταχθούν αυτές οι ουσίες στο παράρτημα 14. Ο συνάδελφος, ευχαριστώ. Καταρχήν ως προς τη διεθνή πτυχή που εφήγει, νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση από την Επιτροπή, αν και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ντάνσετ θα προσθέσει τη δική του οπτική από πλευράς Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών και να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, γιατί υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε κάνει με ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα στον κόσμο του Ρίτς. Το Ρίτς είναι κάτι το μοναδικό παγκοσμίως. Και εάν ακούσουμε δηλώσεις του Επιτρόπου μου εδώ ή και αλλού, πολύ συχνά λέει ότι με το REACH φτάσαμε σε μία βάση γνώσεων ως προς τις χημικές ουσίες για να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και εδώ δεν μιλά μόνο συλλογή δεδομένων ε, στο ε, ιστότοπο, μιλά για τη χρήση αυτών των δεδομένων. Οι χημικές βιομηχανίες θα ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για λόγους ασφάλειας και έτσι θα έχουμε αυτό το σχετικό πλεονέκτημα εκτός Ευρώπης και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν αυτή τη νομοθετική οδό, αλλά μετά από εμάς. Και θα συμβαδίζουν ε, ίσως με εμάς, ίσως να μην είναι βεβαίως τόσο φιλόδοξοι όσο εμείς, αλλά θα κινηθούν σε παρόμοιες κατευθύνσεις. Ε, κάτι άλλο τώρα που ανέφερε ο κύριος Ποτότσνικ, ο επίτροπός μου, είναι ότι φτάσαμε στο μεγάλο ακρογωνιαίο λίθο, δηλαδή εφαρμόσαμε το ρίτς για να είμαστε σίγουροι ότι διασφαλίζουμε ε, αυτά τα, αυτές τις ουσίες ως προς ε, το σκέλος της ασφάλειας και τώρα κάνουμε το δεύτερο άλμα στον κόσμο του ρίτς, δηλαδή η Κομισιόν, ο οργανισμός, τα κράτη-μέλη, οι αρχές των κρατών μελών και όσοι εργάζονται σε, ε, άλλα, ως προς άλλα θέματα, απόβλητα, IPPC και ούτω καθεξής, ενδιαφέρονται για την ε, χρήση αυτών των πληροφοριών για τις χημικές ε, ουσίες για να δουν κατά πόσο είναι χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες για τους παρασκευαστές και για τους εισαγωγείς αλλά και για μας τους ίδιους για να φτάσουμε στους στόχους μας και στους ε, στόχους του Ρίο 20, αλλά βάση περιπτώσει τους στόχους του 2020 στη διάσκεψη, όπως ορίστηκαν στη διάσκεψη κορυφής για την βιώσιμη ανάπτυξη έτσι ώστε να εφαρμοστεί ανά τον κόσμο αυτό το πλαίσιο για την μείωση των κινδύνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ε, Νομίζω ότι έχετε πολλές ερωτήσεις τις οποίες να απαντήσετε, κύριε Διευθυντά. Μερικές από αυτές ίσως επεκτείνονται πέραν των αρμοδιοτήτων του οργανισμού σας, διότι Υπάρχουν και θέματα που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο ή το ρυθμιστικό που ίσως δεν σας αφορούν άμεσα. Αλλά όταν δούμε τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Χημικής Βιομηχανίας βλέπουμε ότι είναι εξαιρετικά. Αυτό είναι ένα ε, παράδειγμα πολύ καλής ρύθμισης. Βοηθήσαμε και στον τομέα της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων πρόκειται για ε, μία ρύθμιση που αφορά την βιωσιμότητα των ε, επιχειρήσεών μας. Κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, διατηρούμε πάντα την ισορροπία των διαφόρων στόχων έναντι το Ριτ και πάντα σε προοπτική σχέση με τις δικέ μας αντιδράσει. Θα ξεκινήσω όμως με το ζήτημα τη αξιολόγηση και τι σχετικέ ερωτήσει. Θα ήθελα να κρατήσω καταρχά σαφέ ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή δεν διαθέτουμε, δεν έχουμε ξεκάθαρη ιδέα ω προς την αναλογία φακέλων που βρίσκεται το 2010 και που ήταν ανεπαρκής ως προς την ποιότητα, ήταν ατελής. Θα πρέπει να σας εξηγήσω ότι το πρώτο αυτό χρόνο, τα πρώτα χρόνια κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταγράψουμε τις ε, καταχωρήσεις των πρώτων ετών, να τις αξιολογήσουμε, να βεβαιωθούμε ότι ότι είναι ικανοποιητική η ποιότητά τους. Έτσι λοιπόν εξετάζουμε περισσότερο τους φακέλους εκείνους των οποίων η ποιότητα δεν ήταν επαρκή. Τώρα μόνο μπορούμε να στραφούμε έχοντας πια λάβει την ε, πλειονότητα των φακέλων, και όταν έχουμε δει την πλειονότητα ε, μαζί με τους τελευταίους φακέλους που κατατέθηκαν πριν το πέρας της ε, προθεσμίας μπορούμε να έχουμε μια εικόνα της ποιότητας τους κατά μεσόρων. Αλλά όχι τώρα. Βεβαίω. Εάν είναι ατελεί οι φάκελοι, πάντα αναλαμβάνουμε δράση. Αν ε, δεν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης, να κάποια μέτρα ή αλλιώς στέλνουμε μια επιστολή ε, όπου ζητούμε βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών από την επιχείρηση και σας διαβεβαιώ ότι οι αποφάσεις αυτές αποστέλλονται και για επαλήθευση στα κράτη-μέλη και στη συνέχεια τη Σχετική Επιτροπή των Κρατών Μελών, όπου κάθε δύο μήνες οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν περί τα 10, 12 και περισσότερα ε, πακέτα, φακέλους δηλαδή, ε, ταυτόχρονα για να βεβαιωθούν ότι πληρούνται εξίσου οι υποχρεώσεις για πληροφόρηση. Άρα η προειδοποίηση αυτή πάει και στην επιχείρηση αλλά και στις αρχές, αρχές αρμόδιες για την επιθεώρηση που μπορούν να επαληθεύσουν οι ίδιες την έλλειψη ή την πληρότητα δηλαδή των ε, πληροφοριών που διατίθενται. και από πλευρά μα επίση επαληθεύουμε και αν δεν είναι πλήρε πληροφορίε, ενημερώνουμε τι σχετικέ αρχέ επιθεώρηση των κρατών μελών που αναλαμβάνουν, εάν χρειάζεται, μέτρα. Ταυτόχρονα, αλλά και, και εμεί κοιτάμε αν έχουμε αρμοδιότητα για να ανάληψη κάποιε δράσει ή απόφαση. Άρα δεν μπορεί κανεί να ξεγλιστρήσει εύκολα. Τώρα αν πρέπει να ανεβάσουμε το ποσοστό μα πάνω από το 5% είναι κάτι το οποίο βλέπουμε σαν προοπτική μακροπρόθεσμη. Αλλά πάντως το 5% είναι ο στόχος μας για οτιδήποτε καταχωρίζεται ε, μέχρι το 2013. Και μετά, από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε υψηλότερο ποσοστό και για τους καταχωρημένους φακέλους. Γιατί δεν περιμένουμε στην επόμενη προθεσμία για καταχώρηση τόσο μεγάλο αριθμό ε, καταχωρήσεων, προτάσεων για καταχώρηση. Δεν σταματάμε δηλαδή το 2013 την καταχώρηση των φακερών. συνεχίζουμε και μετά. φάκελοι, μικροφάκελοι που έχουν κατευθεί πριν από την προθεσμία. Έχουμε ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, επιχειρήσεις που μας έχουν δώσει στοιχεία και σε ποιο σημείο ο φάκελος, σε ποιο σημείο κοινοποίηση αφορά επικίνδυνες ουσίες. Έχουμε ενημερώσει λοιπόν εκτεταμένα την Επιτροπή και πιστεύω ότι και η Επιτροπή θα σας παρουσιάσει έκθεση σχετική αργότερα μέσα στο έτος, έτσι ώστε να σας στηρίξει και στην έκθεσή σας. Συνεχίζεται λοιπόν η αξιολόγηση. Υποχρέωση για καταχώρηση. Όπως είπε η κυρία, μάλλον τέλη καταχώρησης ή επιβάρυνση, άχθος καταχώρησης, όπως είπε η κυρία Γκρόστετ, είναι μάλλον βαρύ το άχθος για ορισμένε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχει αναγνωριστεί και από τα κράτη-μέλη ότι είναι μεγάλο το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το άχθος καταχώρησε, αντιλαμβανόμαστε φυσικά και εμείς τη διάσταση αυτή και ε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επικρίσεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο μέγιστο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το καθήκον αυτό που έχουν να επιτελέσουν και ιδιαίτερως ήθελα να υπενθυμίσω ότι έχουν θεσπιστεί οι θηρίδες στήριξης, τα help desk όπως ονομάζονται από τα κράτη-μέλη, εθνικά help που και εμεί όμω στηρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει όμω η δουλειά του είναι να προσφέρουν στη γλώσσα τη χώρα ενημέρωση μικρομεσαίε επιχειρήσει, ακόμη και κατάρτιση, ακόμη και ε, ενεργό υποστήριξη, αρρωγή δηλαδή όταν συμπληρώνουν του φακέρου στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η σχετική γνώση από πλευρά τη επιχείρηση που θα καταχωρήσει προϊόντα, ακόμα και ένα μικρομεσαίες επιχείρηση πρέπει να έχει τι σχετικέ τεχνικές γνώσεις σε τελευταία ανάλυση απαιτείται να έχει, γιατί αν αγοράζει κανείς από έναν προμηθευτή μια χημική ουσία, πρέπει να γνωρίζει ο προμηθευτής τι πολύ θα ήταν μάλλον κακό να απολύτε κάτι το οποίο μπορεί να είναι ενδεχομένω επικίνδυνη ουσία και πολύ επικίνδυνη ουσία χωρί τι τεχνικέ γνώσει να τι διαθέτει αυτό που πολύ αγοράζει. Εν λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που βλέπουμε σε ορισμένα κράτη-μέλη ότι λαμβάνουν δηλαδή υπόψη το γεγονό ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει χρειάζονται και συμβούλου, Φερρυπίν, που θα παρακολουθήσουν, θα προετοιμάσουν του ε, φακέλου. Ορισμένε χώρε έχουν προσφέρει, έχουν ετοιμάσει συστήματα ε, υποστήριξη και στη χρηματοδότηση ακόμη για τους ε, συμβούλους. Από την άλλη, Πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακολουθούν λίγο πολύ την πορεία των ηγετικών επιχειρήσεων και στο τέλος ε, εξαγοράζουν την επιστολή ε, που αφορά την περιγραφή των χημικών τους και άρα εν τέλει η δουλειά που τις επιβαρύνει είναι μάλλον περιορισμένη και μπορούν να συμμετέχουν με περιορισμένο μάλλον κόστος ε, στη διαδικασία. Βέβαια πρέπει και αυτές από πλευρά να καταβάλουν ε, το σχετικό, τη σχετική επιβάρυνση. Δεν μπορούν βέβαια να αποφύγουν το κόστος της επιστολής πρόσβασης. και Εξήγησε νομίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι αξία μπορεί να έχει και σε ανταγωνιστικού όρου, στο διεθνή δηλαδή, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα μια επιχειρήση, η ποιότητα των πληροφοριών που θα περιλαμβάνονται στη σχετική επιστολή, το να γνωρίζει δηλαδή η επιχείρηση πώ μπορεί να αξιοποιεί, να χρησιμοποιεί κατά τρόπο ασφαλή τι ε, χημικές ουσίες και κυρίως να είναι σε θέση να εξηγεί στον επόμενο χρήστη, στον αγοραστή δηλαδή ή τον μεταποιητή στη συνέχεια, την ασφαλή χρήση αυτών των ουσιών. Άρα θέλουμε να έχουμε στο δυνατόν πιο καλή καταχώρηση. Εγώ προσωπικώς απευθύνω έκκληση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που το επιθυμούν να καταγράφονται και να ε, τις παρακολουθούμε κατά αυτόν τον τρόπο ως προς την ε, τις ανάγκες τους, ε, την ανάγκη για βελτίωση της καταχώρησης. Αυτό θα μας βοηθήσει και εμάς βέβαια για να βελτιώσουμε την καταχώρησή μας, να βελτιώσουμε την καταχώρησή μας μετά το 2013 και χρειάζεται συμμετοχή των ενωτών περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαδικασία αυτή που θα μας βοηθήσει όπως είπα ιδιαίτερως. για δέτη τα εθέρια έλαια μάλλον θα μας απασχολήσουν το 2018 γιατί αφορούν τους μικρότερους όγκους. Ε, επίσης, ε, τεχνική πραγματογνωμοσύνη. Νομίζω ότι δεν υπάρχει επαρκής τόσο στις μεγάλες όσο και στις ε, μικρότερες επιχειρήσεις. Υπάρχει σπάνης εμπειρογνωμόνων ικανών να αξιολογήσουν τις ουσίες αυτές και γι' αυτό ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επιτροπός Ταλιάνη, μας ζήτησε να προσφέρουμε ισχυρά βοηθείες και έτσι ετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα πτυχίου που θα επιτρέψει στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα να συμπράξουν, να συνεργαστούν και να εξασφαλίσουν ε, κατάρτιση για τους επιστήμονες και στην νομοθετική, ε, στην νομοθετική πλευρά της επιστήμης, αλλά και στην κατάρτιση που χρειάζεται για την ε, στοιχειοθέτηση ενός φακέλου υπό τον κορονισμό Ρίτς. Αυτό νομίζω είναι και ο κύριος ε, Πρόντι. Επίσης μίλησε ο κύριος Πρόντι για την ανάγκη να υπάρχει μια ε, κοινή ορολογία που θα χρησιμοποιούν οι νομοθέτες αφενός οι επιστημονικές ε, οι ομάδες επιστημόνων αφετέρου ως προς το τι ε, αντιμετωπίζουν έχει αντιληφθεί νομίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάσταση και ως εκ τούτου έχει ζητήσει με την ε, Γενική Διεύθυνση για την Υγεία των Καταναλωτών Επικεφαλής την ε, διεξαγωγή περισσότερων και τακτικών συναντήσεων μεταξύ αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των νομοθετικών οργάνων των αρμόδιων επασπιτός για την νομοθετική πρόταση έτσι ώστε να γίνεται και αξιολόγηση του κινδύνου κατά τρόπο πιο ξεκάθαρο, με γλώσσα πιο κοινή. Επίσης, ε, καταρτίζουμε, στοιχειοδοτούμε μάλλον μια βιβλιοθήκη για την αξιολόγηση του κινδύνου σε όλες τις γλώσσες, Εναρμονίζουμε δηλαδή, όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά ταυτόχρονα μπορούμε να διατυπώσουμε όλες αυτές τις έννοιες, τις σχετικές με την ασφάλεια στη χρήση των χημικών, σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρη στην προσπάθεια που έχουμε αναπτύξει. Και είναι και αυτό σημαντικό. Για να επανέλθω τώρα στην κυρία Κλάς και τα σχόλιά της. Ιδιαίτερα ως προς τα τέλη. Ναι, το όντι, το ρίτς μερικές φορές προβλέπει τέλη που μπορεί να αποδειχθούν πολύ ψηλά πρόσκομα. Γιατί ιδιαίτερος, διότι οι επιχειρήσεις ε, καταβάλουν, προκατα... μάλλον προκαταβάλουν κατά τη στιγμή της καταχώρησης για όλο το ε, παρεπόμενο έργο που θα επιτελέσουμε εμείς, ε, την αξιολόγηση δηλαδή, του φακέλου, την αξιολόγηση των ουσιών, και σε ένα βαθμό και το έργο αξιολόγηση κινδύνου. Πάλι από τα ίδια τέλη χρηματοδοτείται. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσείς θα αποφασίσετε. Είναι ίσως αμφισβητήσιμο. Η ε, ελέγχεται η σκοπιμότητά του. Εσείς θα αποφασίσετε όμως τι είδους αιτήσια τέλη θα πρέπει να ζητούνται και να μειώσετε ενδεχομένω σημαντικά το κόστος αυτό ή να ζητείτε την προκαταβολή των ε, τελών αυτών ε, με την επιφύλαξη ότι στη συνέχεια θα υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιούνται με προσοχή και κατά τρόπο ασφαλή τα κονδύλια αυτά, έτσι ώστε να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε όπω γίνεται τώρα στην περίπτωση του ΡΙΤΣ για περισσότερα χρόνια τη δική μα δουλειά. Αλλά όπω είπα, εσεί ω νομοθέτε θα πρέπει να κοιτάξετε ε, τα υπέρ και τα κατάνοστα του συστήματο. Για δε τι συνεργατικέ σχέσει μεταξύ βιοκτώνων, μεταξύ νομοθεσία περί βιοκτώνων και Ρίτ. Εμείς ήδη προσπαθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό να αναπτύξουμε αυτές τις, ε, αυτούς τους συσχετισμούς, αυτές τις συνεργατικές σχέσεις και πάνω απ' όλα προσπαθούμε να έχουμε ε, εργαλεία πληροφορικής χρήσιμα τόσο για τον επιστήμονα όσο και, για την επιχείρηση, τόσο για την καταχώρηση και για την αξιολόγηση κινδύνου, για την ενημέρωση ε, που κομίζουμε από την καταχώρηση ή σε μια άλλη περίπτωση από την αδειοδότηση, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτές οι πληροφορίες να αξιοποιούνται από τον επόμενο χρήστη στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό ακριβώς αξιοποιούμε τώρα, προσπαθούμε να ετοιμαστούμε και συνεχίζουμε τη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει κόστος προς την αδειοδότηση των βιοκτώνων, γιατί πάλι υπάρχει κόστος ή τέλος σχετικό με τη διαχείριση των φακέλων, τη γραφειοκρατική δηλαδή διαχείριση. Από την άλλη, το γενικότερο κόστος προσπαθούμε εμείς να το ε, ε, ε, ελαχιστοποιήσουμε χάρη σε αυτές τις, τις συνεργατικές που ανέφερα σχέσεις. Βέβαια, εσείς μας λέτε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια ε, ουσιαστική απόδοση λογαριασμών ως προς το τι έχουμε δαπανίσει για την, πτυχή, για την πτυχή των βιοκτώνων και τι για την αδειοδότηση του ΡΙΤΣ. Για να γνωρίσετε τι είδου ε, τέλη του ΡΙΤΣ μπορεί να αξιοποιηθούν για τα βιοκτώνα. Άρα καταγράφουμε ως μήνυμα ότι θέλετε από πλευράς μας μια ε, επακριβή αξιολόγηση της ε, κατανομής του κόστους και για τα διοκτώμενα, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι ήδη πράττουμε. Επίσης πιστεύω, αλλά δεν έχω ακριβή στοιχεία για τα τέλη. Πιστεύω όμως ότι αντίστοιχες ε, μειώσεις στην επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε πρόκειται για μικροεπιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, υπάρχει σημαντική έκπτωση από τα τέλη που καταβάλουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και θα ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι έχουμε πράξη τέλη καταχώρησης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μας επιτρέπουν αυτές ε, οι προεισπράξεις να, να λειτουργούμε και να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του κανονισμού REACH στον ε, αιώνα των άπαντα. Το 2014 θα έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια αυτά που έχουμε προεισπράξει και άρα θα πρέπει να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση του νομοθέτη, δηλαδή την μεικτή τη συγχρηματοδότηση, τη μεικτή χρηματοδότηση, δηλαδή εν μέρη από τα τέλη και εν μέρη από επιδοτήσεις, το καθεστώς δηλαδή εκείνο το οποίο θα ε, μας επιτρέψει να περάσουμε το προσοχές δημοσιονομικό πλαίσιο και ελπίζω όταν έρθει η ώρα να εξετάσετε το προσοχές δημοσιονομικό πλαίσιο να το έχετε και αυτό υπόψη. Κατάλογος υποψηφίων. Ναι, έχουμε ήδη την ε, ιδέα αυτή και ιδιαίτερα το στόχο για όλους μας και ένα κατάλογο για 130 ουσίες για τον επόμενο χρόνο. αλλά προσπαθούμε και εμεί βέβαια και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να είμαστε έτοιμοι του επόμενου μήνε στη δουλειά που έχουμε να κάνουμε. Προσπαθούμε δηλαδή εμεί από πλευρά μα να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη, γιατί βεβαίω είναι διατεθειμένα να ε, συμμετάσχουν σε αυτή τη δουλειά και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πρώτη συνεδρίαση προγραμματισμού, όπως προβλέπετε, στα τέλη του έτους στην υπηρεσία μας όπου θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα κανονισμό που θα καθιστά όχι μόνο εμά και την Επιτροπή υπεύθυνου για τον προσδιορισμό ε, στόχων, αλλά ε, και τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι έτσι έχω απαντήσει, ελπίζω τουλάχιστον, ότι έχω απαντήσει. βέβαια πολλά ακόμα. Ε, ενημερωνόμαστε, παίρνουμε το feedback όπως λέμε από τις υπηρεσίες. Στη προσπάθεια για τις ε, γλώσσες και για να είμαστε έτοιμοι στο βέλτιστο δυνατό βαθμό. Κύριος Ντέιβις. Μια ερώτησή μου όμως δεν απαντήθηκε. Μπορείτε να μας πείτε πώς αξιολογείτε την ανταγωνιστική θέση της χημικής ε, της Ευρώπης ε, μετά το ρίτσο έχει βελτιωθεί, έχει... είναι σε δυσμενέστερη θέση ή είναι στην ίδια κατάσταση όπως Ευχαριστώ. Φυσικά νομίζω ότι αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει αυτό το θέμα, γιατί εκείνοι μελετούν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η βιομηχανία και έχουν αρχίσει και μελέτες. Ελπίζω του χρόνου να είναι η Επιτροπή σε θέση να απαντήσει, διότι θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες. Από, από αυτά που βλέπω εγώ, αυτή τη χρονική στιγμή Φαίνεται ότι ένας πάρα πολύ μεγάλος ε, συντριπτικός αριθμός επιχειρήσεων κατόρθωσε να υποβάλει την, ε, να εγγραφεί στο Μητρό κυρίως ε, στην επωνομαζόμενη downstream βιομηχανία, δηλαδή στα τέλη της βιομηχανικής αλυσίδας. δηλαδή θα, δεν είναι εκείνοι που επηρεάζονται αν θέλετε πρώτοι από την έλλειψη κάποιων χημικών ουσιών, μάλλον στην αρχή της αλυσίδας ε, επηρεάζεται η βιομηχανία. Επίσης υπάρχει ομάδα ε, όπου εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Βιομηχανία και ο οργανισμός μας ε, και η Επιτροπή μας δεν έχει διαπιστώσει κάποιο τέτοιο κρούσμα Γι' αυτό κρίνω πως είναι σε θέση να ανταγωνιστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία, έχοντας βέβαια υπομειστεί ήδη το κόστος της πρώτης ε, καταχώρησης. Αυτό πιστεύω αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Νομίζω, κύριε Διευθυντά, ότι από απαντήσατε διεξοδικά σε όλες τις ερωτήσεις. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε τον οργανισμό σας. Σας ευχαριστούμε για αυτό τον απολογισμό, την έκθεση που μας παρουσιάσατε. Είναι πολύ θετικά τα πορίσματα και προτείνω να περάσουμε στο σημείο 6 της μερικής διάταξης. Πρόκειται για μία ερώτηση για τον ιό HIV. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση για την καταπολέμηση του AIDS στην Ευρώπη και στις γειτονικέ χώρες για την περίοδο μέχρι το 2013 και η πολιτική είχε επικεντρωθεί σε τρία βασικά σημεία δεν υλοποιήθηκαν αυτά που είχαμε προβλέψει και αυτά που επιθυμούσαμε, εξού και η προφορική ερώτηση. Δεν ξέρω ποιος από τους συνυποβάλλοντες θα, το, ήθελε το λόγο, η κυρία Γκροστέτ, κυρία Σίλντερς, για να μας παρουσιάσετε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη λέει η κυρία Γκροστέτ. Ε, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό που ασχολούμαστε με αυτό το ερώτημα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει τις δυσάρεστες ε, διαπιστώσεις τωρινής κατάστασης, ε, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Το Νοέμβριο 2008 το ψήφισμά μας ζητούσε πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή. Αυτό το ψήφι... Μετά από αυτό το ψήφισμα ακολούθησε και μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την καταπολέμηση του HIV στην Ευρώπη και στι ε, γειτονικέ χώρε για την περίοδο 2009-2013 και ένα σχέδιο δράση για να μειωθεί ο αριθμό των νέων κρουσμάτων HIV. Το είπατε όμω Πρόεδρε, δεν έχει σημειωθεί ιδιαίτερη πρόοδος και παρατηρούνται νέα κρούσματα και στην Ευρώπη και στι γειτονικέ χώρε. Δεν μειώνει το αριθμό των κρουσμάτων και βάσει τη αποτίμησης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψη και Ελέγχου των Νόσων 30% των οροθετικών στην Ευρώπη κατά μέσο όρο δεν έχουν είναι διαγνωστεί ω τέτοιοι ε, και άρα δεν γνωρίζουν ότι έχουν μολυνθεί από τον ιό ε, HIV ε, και άρα ο κίνδυνος μετάδοσης του HIV είναι κατά 3,5 φορές υψηλότερη σε σχέση με κάποιον που έχει διαγνωστεί. Οι οροθετικοί λοιπόν θεραπεύονται με μεγάλη καθυστέρηση και λόγω αυτού έχουν φτάσει σε προκεχωρημένα στάδια μόλυνση πρωτού καν γίνει η διάγνωση πόσο μάλλον αρχίσει η θεραπευτική αγωγή. Η μελέτες μας επιτρέπουν να ανασχεδιάζουμε και να επανεξετάζουμε την πολιτική αντιμετώπιση του HIV. Έχει αποδειχθεί, παραδείγματο χάρη, ότι ένα οροθετικό ε, που παίρνει ε, τα ρετροϊκά φάρμακα μετά τη διάγνωση νωρίτερα, πριν αρχίσει να εκφυλίζεται η υγεία του, ε, μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο διάδοση του ιού σε μη μολυσμένου σεξουαλικού συντρόφου, παραδείγματο χάρη. Βλέπετε τη σημασία τη διάγνωση, τη πρόληψη χρειαζόμαστε πρόορη πρόληψη και πρώιμη θεραπευτική αγωγή στην Ευρώπη. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να δαμάσουμε αυτήν την ε, νόσο. Ε, βρισκόμαστε στα μέσα περίπου του σχεδίου δράσης και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσουν μεγαλύτερη προσοχή την πολιτική πρόληψη υπό το φως των νέων εξελίξεων και των νέων στοιχείων σε σχέση με την πρόσβαση στην ε, διάγνωση του κοινού και θα πρέπει να υλοποιήσουν όλα τα μέτρα για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που στην στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το έτσι στη Νέα Υόρκη πέρσι τον Ιούνιο. Ε, αποτελεσματική δράση κατά του HIV στις ε, περιφέρειες προτεραιότητας, στις περιοχές προτεραιότητας και επίσης να βρούμε τις πληθυσμιακές ομάδες που είναι ε, οι πλέον ευάλωτες για τον ιό αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι δύο στόχοι νομίζω απαιτούν μια ιδιαίτερη δραστήρια πολιτική από πλευράς μας και αυτή είναι και η σημασία, η ουσία της ερώτησής μας. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτη. Κυρία Σίλτερς τώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια στην ιατρική περίθαλψη. Έχει σημειωθεί πρόοδος και ξαφνικά χαλαρώσαμε, αν θέλετε, όλοι με αυτόν τον ιό HIV. Προσοχή λοιπόν, γιατί έχουμε φτάσει στα μισά του δρόμου. να αρχίσουμε να καρκινοβατούμε τώρα στην πολιτική πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών, όπως το HIV-AIDS. Υπάρχουν διάφοροι τομείς που πρέπει να μας απασχολήσουν όλους ιδιαίτερως ε, μέσα στο ψήφισμα. Παραδείγματο χάρη οι πληθυσμιακές ομάδες που συνιστούν προτεραιότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν σωστές αποτιμήσεις και πιο στοχοθετημένες εκστρατείες ενημέρωσης, ώστε να προστατεύσουμε συγκεκριμένα αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες. Επίσης, ε, οι πολιτικές και τα σχέδια δράσης θα πρέπει ε, φυσικά να συνάδουν με τις πολιτικές ε, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όμως στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να καθοδηγούμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας έχοντας ε, κατά ότι θα πρέπει να παραβιάζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, όσων έχουν προσβληθεί από αυτόν τον ιό και μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για ευάλωτες κοινότητες ε, και θα έπρεπε να προωθήσουμε και πολιτικές αξιολόγησης και να εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση και στη διάγνωση και στην θεραπευτική αγωγή χωρίς καμία, κανένα περιορισμό. Επίσης να διαλύσουμε αυτούς τους μύθους για, τους, για όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό χρειαζόμαστε τη ευρύτατη υποστήριξη από διασημότητες, από πολιτικούς καθώς και επαρκή κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι θα προωθήσουμε την ενημέρωση του κοινού. Ε, η πρόληψη λοιπόν για τις βασικές ε, ομάδες ε, και για τις βασικές περιοχές που πλήττονται από τον ιό αυτό είναι το κεντρικότερο στοιχείο σε μια μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς στον 21ο αιώνα παραμένει το AIDS μια από τις βασικότερες απειλέ για τη δημόσια υγεία. Ευχαριστούμε. Ο Κρίς Ντέιβις έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Τον Παβανόβα είναι σκιώδης εισηγήτρια, δεν είναι εδώ, καθυστέρησε και μου ζήτησε να αναφέρω τα εξής. Η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει το σχέδιο ψηφίσματος, καλωσορίζει τις προτάσεις για την πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή, για την ε, πρόορη ε, ε, διάγνωση και πρόορη θεραπεία. Επίσης, ναι, επικεντρώνει το ενδιαφέρον στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για, την, για τον έλεγχο της νόσου στην Ένωση και στις γειτονικές χώρες Βέβαια θα δούμε αν συμφωνούν οι συνάδελφοι και αν διαφωνούν ως προς τη φρασιολογία δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να το διαπραγματευτούμε επίσης. πιστεύει ότι ε, πρέπει να προωθήσουμε τις ε, εκστρατείες ευαισθητοποίησης ε, κυρίως για τους ομοφιλόφιλους, για τους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών, δηλαδή τις πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Επίσης να καταπολεμήσουμε το στίγμα που φέρουν αυτοί οι άνθρωποι στα μάτια των υπολείπων. Ε, χρειάζεται μια αποτίμηση των εφιστάμενων πολιτικών καταπολέμησης και πρόληψης του HIV και σε σχέση με τους ε, κινδύνους και τις ανησυχίες διάδοσης ε, της νόσου σε γειτονικέ χώρες. Νομίζω ότι χρειάζεται μια επαναξιολόγηση των πολιτικών μας. Τέλος, είναι η Αντωνία Παβανόβα, τονίζει ότι δίνουμε, είμαστε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους μεγαλύτερους δωρητές στα προγράμματα καταπολέμησης της νόσου και άρα χρειαζόμαστε μία παράγραφο μέσα στο ψήφισμα ε, όπου θα εξηγούμε με ποιο τρόπο συλλογικά και σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους πόρους που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον έλεγχο της αρρώστιας. Bien, je vous remercie. Alors, je crois qu'il n'y a... Σας ευχαριστούμε και δεν ζητάει κανείς άλλο στο λόγο για αυτό το θέμα. Οπότε θα στήσω από τον κύριο Έμπελ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Παρακαλούμε. Σας ευχαριστούμε και θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί έχουμε καθυστερήσει. Είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα και έχει ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή να κάνει αυτή την πολιτική δήλωση για την αντιμετώπιση του AIDS. Ε, αυτό είναι το κλειδί. Και ούτως ή άλλως αυτό το στοιχείο είναι και στον πυρήνα της πολιτικής μας θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Θα... Είμαι σύντομος. Πρώτον και σε σχέση με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα, έχουμε δύο παράλληλες και αλληλένδετες πολιτικές, δηλαδή η πολιτική αντιμετώπιση του HIV στα κράτη-μέλη της Ένωσης και στις γειτονικές χώρες και μια άλλη στρατηγική σε διεθνές επίπεδο σημειώνονται εξελίξεις και στα πλαίσια, στα πλαίσια και των δύο πολιτικών και καλό θα ήταν να δούμε αν ε, συμβαδίζουν αυτές οι δύο πολιτικές. Δεύτερον, ε, αν έχει σημειωθεί πρόοδος στο συντονισμό της δράσης ε, των κρατών μελών, της κοινωνίας των πολιτών, όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τόσο ώστε κάποιες περιοχές και κάποιες πληθυσμιακές ομάδες να αναδειχθούν σε προτεραιότητα και νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής. Χρειάζεται καλύτερη στοχοθέτηση της μας και έτσι επιτυγχάνουμε και προβολή των προσπαθειών που κάνουμε σε αυτό το τόσο σημαντικό τομέα τρίτον σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και πρόληψη ε, των Νόσων έχουμε ήδη μία έκθεση παρακολούθηση. Ε, βλέπουμε κατά πόσο υλοποιούνται οι δεσμεύσει ε, των κρατών μελών και μέσω τη διάσκεψη του Δουβλίνου βλέπουμε κατά πόσο εφαρμόζει τι δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και πρόληψη. έχουμε ήδη στη διάθεσή μα στοιχεία για το πρώτο ήμιση του σχεδίου δράσεω και έχουμε τα απαιτούμενα εφόδια για να δούμε δεδομένο των εξελίξεων πώς θα πρέπει να κινηθούμε κατά το δεύτερο ήμιση του σχεδίου δράσης. Πρόεδρος, μάλιστα σας ευχαριστούμε. Έχουμε εδώ πέρα τον ε, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Όσων, τον κύριο Σπρέγγερ. Σίγουρα έχετε πολλά να μας πείτε για αυτό το θέμα, οπότε θα θέλαμε να σας ακούσουμε. Παρακαλώ. Ε, e Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε τελικανοποιημένοι για το ότι χρησιμοποιείτε το υλικό που ετοιμάζουμε εμείς και ότι το χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την χάραξη πολιτικής πάνω απ' όλα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι συμφωνώ ιδιαίτερως με τα όσα υπόθηκαν εδώ. Αλλά, λόγω της οικονομικής κρίσης, ενδέχεται ορισμένε χώρες να μην είναι πάντα διατεθειμένες να δώσουν την ίδια προσοχή στην ε, πρόορη διάγνωση που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και καταγράφεται επίσης ο κίνδυνος αυτός της ε, καθυστερημένης διάγνωσης. Επίσης πολύ σημαντικό είναι όταν διαγνώσκεται κάποιος ε, ως θετικός, να έχει και την κατάλληλη αγωγή στη διάθεσή του. Μην το λησμονείτε αυτό. Καλώς σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να στεί κανείς άλλο στο λόγο. Και υπενθυμίζω ότι έχουμε προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια εγκρίνεται σε επίπεδο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στις 22 Νοεμβρίου η έκθεση και στην Ολομέλεια πάει τον Δεκέμβριο, στην 1η του Δεκεμβρίου. Η σε διάταξη λοιπόν στο επόμενο θέμα τώρα. Ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Μάρκεν Σπέγκερ, Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Παρακαλώ να έρθετε εδώ κοντά μας στο βήμα. Έχετε το λόγο κύριε Σπρέγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να επισημάνω ότι με χαρά καλώς ορίσαμε την κυρία Γιάννα Κουδάκη, την κυρία Αγιούσο, τον κύριο Φέλνερ και πρόεδρο της Επιτροπής ε, τον προηγούμενο μήνα Χρήσιμες λοιπόν όλες τις συζητήσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστώ την, ξεκινώντας μάλλον να ευχαριστώ τη Μαρίνα που είναι εδώ, που δεν είναι εδώ, αλλά για, πάνω απ' όλα θέλω να την ευχαριστώ για τις προσπάθειές της, για την ενέργεια που αφιέρωσε στην ε, υπηρεσία μας και προκαταβολικά θα ήθελα να την ευχαριστήσω για την ε, προσπαθήσει να φιλοξενήσει εκδηλώσεις για λογαριασμό μας. Όταν έλαβα, λοιπόν εγώ ως διευθυντής μου ζήτησε η κυρία Νακιουδάκη να έρθω ως ε, το δυνατόν πιο συχνά στο Κοινοβούλιο και χαίρομαι που υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν στις 22 Νοεμβρίου το μεσημέρι μαζί με την κυρία Κάριν Κάρνμπαχ θα έρθουν σε μια ενημέρωση της, ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για, την, ε, για τον εμβολιασμό ε, κατά της γρήπης. Αν θυμάστε από την περσινή σας έκθεση της κυρίας Ριβαζή, είχα υποσχεθεί ότι θα δώσουμε στις, ε, στα μέλη της Επιτροπής σας ό,τι στοιχεία έχουμε για το πρόγραμμα εμβολιασμών εν ώψη της προσεχούς περίοδου εμβολιασμού. Έτσι λοιπόν ο, συντονισμό, ο συντονιστής ε, κ. Σάγκος μαζί με τη Γενική Διεύθυνση για την Προστασία της Υγείας του Καταναλωτή και ο φαινόμενο σα κάνω την παρουσίαση τον Νοέμβριο. Στι 30 Νοεμβρίου, κυρία ε, Γιανακουδάκη θα ε, κηρύξει την ημέρα κατά του AIDS ε, που έχει υπό την αιγίδια της. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Φυσικά θα σας προσταρούν οι σχετικές προσκλήσεις. Επίσης σήμερα, ο Γιάννα θα ε, κηρύξει το πέρα των επιστημονικών μας εργασιών στο Κχόλμις 8 Νοεμβρίου και θα ε, τεθεί επικεφαλής του, ε, των εργασιών του Διοικητικού μας Συμβουλίου την επομένη. Θα ήθελα όμως και να αναφερθώ στην επίσκεψη της Στοκχόλμη, στη Στοκχόλμη, της αντιπροσωπείας σας. Πριν όμως περάσω σε αυτό, επιτρέψτε μου να στρέψω την προσοχή μου σε κάτι άλλο Μάλιστα. Ναι, λοιπόν θα πρέπει να, επισημάνω ότι δεν έχω χρηματοδότηση ούτε εγώ ούτε η υπηρεσία μου, το κέντρο πρόληψη δηλαδή, ε, χρηματοδότηση από οποιοδήποτε ε, εμπλεκόμενο ενδιαφερόμενο μέρος, ε, τη βιομηχανική δραστηριότητα κτλ. Τα πάντα λοιπόν αποφασίζονται στο ιστορικό του κέντρου ελέγχου των νόσων με την πραγματογνωμοσύνη και τη βοήθεια των ειδικών που έχουμε που είναι όλοι υποχρεωμένοι σε δήλωση συμφερόντων και βέβαια έχετε τη σχετική καταχώρηση στην Ε, σελίδα μας, στην ιστοσελίδα μας. Τώρα θα ήθελα να περάσω πάλι στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας σας, που άλλωστε θα έχετε δει και τις φωτογραφίες. Η αντιπροσωπεία σας έλαβε μέρος στην καθημερινή μας δουλειά, στη δουλειά δηλαδή της ε, επιτήρησης και νομίζω ότι μπορείτε να δείτε από τις πρώτες ε, φωτογραφίες ότι είχαμε κέντρα παρακολούθησης ε, των ε, ε, δηλώσεων επιδημιών, ανακοινώσεων προβλημάτων και το καθεξής ανά τον κόσμο με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ανταπόκρισης το οποίο οργανώνουμε από κοινού με την DG Sanko και έτσι συνδέουμε το εθνικό με το ευρωπαϊκό επίπεδο και τις σχετικές αρχές. Τα κράτη-μέλη αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές και ενημερώνουν τις υπηρεσίες μας. Και έχουμε και μια επιδημολογική ενημέρωση για την φύση αυτών των ζητημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός ε, υγεία αλλά και άλλοι εταίροι ανά τον κόσμο επίση εμπλέκονται στην ενημέρωση, αλλά έχουμε και ανεπίσημη ενημέρωση από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Παραδείγματι, παρακολουθούμε τακτικά σε όλε τι χώρε μέλη. Και έτσι κάθε μέρα, 11 και 30, όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε επίσημα ή ανεπίσημα, συγκεντρώνονται στο χώρο των συζητήσεών μας, τη διαβούλευση, των διαβουλεύσεων και λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. Στις 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν οι πραγματογνωμόνα και οι ε, μελέτησε τα στοιχεία που έχουμε για, τις εξή για τα εξή κρούσματα. Έχουμε ε, την όσο των λιγιοναρίων μεταξύ τουριστών ε, στην, σε ένα στο χωριό της Λαζίζα. Μετά έχουμε περίπτωση ελονοσία σε δύο περιοχές της Ελλάδας με μονομένα κρούσματα και μαγουλάδες στην Ευρώπη που επανεμφανίζονται και ουσιαστικά αφορούν όλα τα κράτη-μέλη. Τρεις λοιπόν απειλές για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε να προβούμε σε μια ταχεία αξιολόγηση κινδύνου. Βλέπετε επίσης ε, τον... Ε, τη διαφάνεια και την υποχρέωση να προσφέρουμε στοιχεία και ενημέρωση ε, στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Τώρα, να σας εξηγήσω λίγο ποια είναι η κίνδυνη. Κοιτάξτε μαζί με, με την αντιπροσωπεία μας όταν μας επισκέφθηκε, με την αντιπροσωπεία σας. Δεν γνωρίζετε τη Λαζίζη, είναι ένα πολύ ωραίο χωριό κοντά σε μια περιοχή της Ιταλίας ε, που έχω επισκεφθεί εγώ προσωπικό είναι πολύ ωραίο χωριό. Οι περισσότεροι τουρίστες που ε, εμφάνισαν τα κρούσματα αυτά ήταν Ολλανδοί και Γερμανοί. Η νόσος των λεγιοναρίων είναι ένα από τα κράτη, από τη, μία από τις νόσους για τις οποίες έχουν ε, τα κράτη-μέλη της με να πληροφορίες για κρούσματα μεταξύ τους αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δώσει λοιπόν τα στοιχεία, έχουμε επισκεφθεί τα ε, Ινστιτούτα και έχουν δοθεί οι σχετικές πληροφορίες βέβαια κατά τρόπο εμπιστευτικό και στη συνέχεια δόθηκαν οι πληροφορίες στους γιατρούς πάλι εμπιστευτικά. Το κέντρο ελέγχου λοιπόν διαπιστώνει με βάση τις πληροφορίες ότι υπήρχαν 7 ε, περιπτώσεις, ε, τα κρούσματα νόσου των λεγεωναρίων ε, από, που εμφανίζονται σε άτομα που είχαν πρόσφατα επισκεφθεί την περιοχή αυτή της Λαζίζα. Το διαπιστώσαμε, βεβαιωθήκαμε και συνέχεια ενημερώσαμε τις Ιταλικές αρχές για την νερολουσία στην Ελλάδα. Και τα άλλα κράτη-μέλη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βεβαίως θέλουν να γνωρίζουν τη σημασία και η διάσταση του φαινομένου ε, υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένω για τουρίστες που επισκέπτονται συγκεκριμένη περιοχή της ε, Ελλάδας. Πρέπει κανείς να αναλάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αποτροπή της επέκτασης της διάδοσης του φαινομένου ή απλώς ε, είναι περιβολικές αντιδράσεις. Είναι τώρα το φαινόμενο αυτό τέτοιο των, ε, της νόστων αυγουλάδων που έχουμε επίσης σαν τρίτο φαινόμενο διαπιστώσει που γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον εξαγωγός κρουσμάτων. Πρόκειται για μια νόσο άκρος μεταδοτική. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν μόνο τους δηλαδή να εξασφαλίσουν ε, απόλυτη προστασία από την μετάδοση της, τη μετάδοση της νόσου. Και θα ήθελα, Πρόεδρε, να ενημερώσω και εσάς και την Επιτροπή για το τι έχουμε κάνει σχέση αυτά τα κρούσματα. Η νόσο των Λεγιοναρίων στην Λαζίζε. Φαίνεται ότι έχει κλείσει, έχει λήξει. Οι Ιταλικές αρχέ ενημερώθηκαν, έλαβαν την τα κατάλληλα μέτρα, ε, εντόπισαν την ε, νόσο αυτή ε, στο σημείο που εφαρμοζόταν στο σύστημα ίδρυυσης και ενημέρωσαν και όποιον άλλο ενδεχομένω είχε εκτεθεί στην στο παράστο. Ε, με ενημέρωση λοιπόν πολύ απλή και ε, ρεαλιστική, γιατί η νόσος μπορεί μόνο με συγκεκριμένο αντιβιωτικό να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν υπάρξει κατάλληλη αγωγή, κινδυνεύει κανείς με πνευμονία, μπορεί να είναι ακόμη και μοιραία. Μόνο χάρη στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, και ενημέρωσης ήταν δυνατή η ενημέρωση και η διάγνωση, η ενημέρωση, η αποτροπή της περαιτέρω επέκτασης του φαινομένου της λόγου των λεγιοναρίων. Για δε την Ελλάδα τώρα έχουμε μια διάδοση περιπτώσεων ελονοσίας 17 εντωμεταξύ σε πέντε διαφορετικές περιοχές. Πριν από λίγες μέρες ε, κατόπιν αιτήματος Ελλάδας ε, δομολόγοι και ειδικοί από την ομάδα μας Πέρασε μια εβδομάδα εκεί για να αξιολογήσουν την κατάσταση και καταγράφουν ότι αυτές οι περιπτώσεις εμφανίζονται σε γεωργικές περιοχές κοντά σε έλλη με πολύ περιορισμένα φαινόμενα τουρισμού. Θα πρέπει να συνεχίσει η Ελλάδα να διαγνώσκει και να ε, προσφέρει την κατάλληλη αγωγή για την ελονοσία, αλλά οι συνέπειες μπορεί να έχει το φαινόμενο αυτό στην, ε, στις υπόλοιπες χώρες είναι πολύ περιορισμένες και έχουμε καταγράψει τις σχετικές μας προτάσεις στην ε, ιστοσελίδα μας που μπορείτε να κοιτάξετε και να συμβουλευτείτε αν το χρειάζεστε. Αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερο όμως είναι η επανεμφάνιση της νόσου των μαγουλάδων. Το αρχές ε, Σεπτεμβρίου είχαμε 26.000 κρούσματα, ενώ τώρα έχουμε φτάσει στις 28.000. Με τρεις επιπλέον θανάτους, συνολικά 10 θανάτους από μαγουλάδες εφέτος. Αυτό νομίζω σημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός τόσο κρουσμάτων όσο και θανάτων μπορεί να ε, έχει υποτιμηθεί. Και ενώ λοιπόν ε, η νόση των στην Ελλάδα, στην ε, Ιταλία και, την, και τις στην Ελλάδα μένουν σε όρια σχετικά λογικά και αποδεκτά, η περίπτωση της παροτίτιδας μας ε, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα Θα πρέπει λοιπόν να ε, μιλήσουμε για την επανοργάνωση και την αποτελεσματικότητα στην επανοργάνωσή μας, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη χρήση και αξιοποίηση του τελευταίου κονδυλίου που διατίθεται σε εμάς. Έχουμε εισαγάγει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό, ένα νέο σύστημα καταγραφή στον προπολογισμό, καταρχάς κοιτάξαμε τι άμεσες δαπάνες, το λεγόμενο τίτλο 3. Ωστόσο τώρα η κατάσταση δεν ήταν ε, Μπορεί να φαίνεται από, τον, ε, από το κατάστοιχο που βλέπετε εδώ ότι δεν υπάρχουν πραγματικά δαπάνες για την ενημέρωση σχετική με επιδημίες. Ωστόσο αυτό δεν, ακριβέ, δεν είναι ακριβές. Το μόνο που διαφοροποιεί την ε, εικόνα είναι ο χρόνος του προσωπικού που αφιερώνεται. Μόνο έτσι μπορεί να καταγραφεί το πραγματικό κόστος των διαφορετικών δραστηριοτήτων για να συστήσουμε ουσιαστικά το πρόγραμμα εργασίας μας. Το Φεβρουάριο ανακοινώθηκε η επανοργάνωση με την Ανδρέα ως υποδιευθύντρια και έτσι έχουμε ε, νέα ισορροπία και βέβαια εκπροσώπηση των φίλων ισομερή. Έχουμε 50% προσωπικό γυναίκες, ωστόσο ε, στη βαθμίδα της διοίκησης ε, το ποσοστό, η παρουσία των γυναικών είναι κάτω από το 40%. Έχουμε όμως προσλάβει μόλις ε, τρία νέα διοικητικά στελέχη, επικεφαλής νομικής υπηρεσίας ε, και επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφορικής. Τρεις και οι τρεις λοιπόν ήταν γυναίκες και βέβαια ήταν και καλύτεροι υποψήφοι. Γι' αυτό προσλήφθηκαν. Για την, για αναδιοργάνωση λοιπόν θα ήθελα να επισημάνω ότι θελήσαμε να προσδιορίσουμε καλύτερα και πιο διαφανώς ε, τις προτεραιότητές μας Έχουμε δύο βασικά ομάδες, δύο ενότητες καλύτερα. Με βάση τις προτεραιότητες της δουλειάς μας έχει γίνει κατανομή των εργασιών και αν αλλάξουν οι προτεραιότητες, εάν εμφανιστεί μια σημαντική επιδημία όπως της ε, νέας γρήπης κτλ, μπορούμε εύκολα να αναθέσουμε τα διαφορετικά νέα καθήκοντα στους ειδικούς μας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε δράση, μακροπρόθεσμη και σχεδιασμό. Ε, των εργασιών μας. Ξέρω ότι έχουν ασκηθεί επικρίσεις κατά του κέντρου μας γιατί δεν είχαμε γιατί παρουσιάσαμε σημαντικές μεταφορές κονδυλίων στον προπολογισμό μας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι ε, ένα από τα κύρια καθήκοντα της ε, υποδικήτριας της κυρίας Ανδρέα Αμών. Είναι δύσκολο βεβαίως, αλλά υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις και βελτιώσεις. Και μόνο 50% του προϋπολογισμού μας θα αντιστοιχεί στις μεταφορές ε, σε σύγκριση με το 27% του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους. Και τώρα για να περάσω στις προτεραιότητες σχετικές με, με τον περιορισμό των δαπανών, Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά σε συνεργασία με τα, στη συνεργασία μας με τα εργαστήρια. Θυμάμαι πολύ καλά ότι ανησυχούσατε, ότι είχατε εκφράσει ανησυχίες ως προς την κίνδυνο της, ε, το, και τα κρούσματα της νέας ε, γρήπης στη Γερμανία. Ένα από τα κύρια, λοιπόν, ε, μια από τις κύριες προκλήσεων ότι τα κρούσματα <clears throat> προξενούσε ένα νέο είδος βακτηριδίου αυτής της ε, της E. coli. Ε, παρακολουθήσαμε την κατάσταση και με ικανοποίηση είδαμε ότι ε, με επικεφαλής των Max Trulens η ομάδα μας, μάλιστα πρόκειται για ένα από τους πιο ικανούς επικεφαλής εργαστηρίων στην Ευρώπη, ανέλαβε να χειριστεί την επιδημία αυτή του E. coli υπήρξε η πρόσβαση για τα εργαστήρια, εξασφαλίστηκε η πρόσβαση για τα εργαστήρια στα σωστά πρωτόκολλα, τη δουλειά δηλαδή την οποία έχουμε να κάνουμε με την ε, Γενική Διεύθυνση για την Προστασία ε, της Υγείας του Καταναλωτού και που θέτει ως κύρια προτεραιότητα την καλή δουλειά των εργαστηριών. Εδώ ε, το ζήτημα του E. συζητείται σε μια διάσκεψη που έχει οργανώσει η κυρία ε, Dagmar ΠΕΡΕΝΤ στις 10 Οκτωβρίου, όπου θα είμαι και εγώ παρόν μαζί με την κυρία Ζησλέα από την ΕΣΑ και με ε, συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Υγείας Κουτραλωτή. Έτσι λοιπόν, και καθώς ξέρω ότι σας απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα της ε, λειτουργίας των κέντρων. Από ποτέ που ανέλαβα τα καθήκοντά μου διευθυντής, επισκέφθηκα σε πολλές χώρες της ε, Ευρώπης τα κέντρα διάγνωσης και πρόληψης ε, λιμοδονώσεων Πήγα στην Ρουμανία Φερρυπίν σε ένα κέντρο υγείας για τους Ρωμά για να αντιληφθώ καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν αυτές οι κοινωνίες και για να αντιληφθώ καλύτερα πώς θα μπορούσε το κέντρο μας να βοηθήσει περισσότερο και τις ομάδες αυτές. Στον κατάλογό σας επίσης θα βλέπετε μια φωτογραφία τριών παιδιών. Είχα πάει και σε ένα νοσοκομείο φυματικών, ε, πράγμα το οποίο μας υπενθυμίζει ότι οι στατιστικές της φυματίας θα πρέπει να κρύβουν τα, την παρουσία πραγματικών ανθρώπων, αυτών που νοσούν από την φυματίωση. Οι προτεραιότητες μας λοιπόν για τον επόμενο χρόνο είναι πολλοί πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ε, εμβολιαστεί κατά κάποια ε, νόσου και αν υπάρχουν πολλοί λοιπόν για κάποια συγκεκριμένη νόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα την ε, κατάσταση. Φερρυπίν στο, στο κρούσμα αυτό της Ιλαράς έγινε μεγάλη προσπάθεια πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας για, την, για τον εμβολιασμό των παιδιών. Θεωρήθηκε, ορίστηκε ως κύρια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητήθηκε η στήριξη και της Γενικής Διεθνή Προσέγγισης του Σχέσου και της ε, δικής μας υπηρεσία. Ο στόχος λοιπόν η προτεραιότητα για το κέντρο το δικό μας θα είναι η εκρίζωση της Ιραράς το 2012. Χρειάζεται βέβαια ε, πολλή δουλειά, αυτό δεν αμφισβητείται, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. 28.000 κρούσματα ηλαράς, όπως είπαμε, έχουν καταγραφεί. Ε, πολύ σημαντικά νούμερα. Και εδώ μπορείτε νομίζω να δείτε, δεν έχει βγει ακόμα στην οθόνη από ό,τι βλέπω, με τα, τις, τα σφαιρίδια που βλέπετε δείχνει ότι ε, δεν έχει ακόμα το θέμα της Σιλαράς ε, ελεγχθεί και δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή, ούτε εμφανίζεται μόνο στο βορρά ή μόνο στο νότο, μόνο στο Ανατολή, μόνο στη Δύση. Έχουμε πολλούς, πολύ μεγάλο κίνδυνο ε, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει και να αναλυφθούν μέτρα και να επιδειχθεί ηγετική ε, στάση. Αυτό σημαίνει παρουσία και του υπεύθυνου υγείας και του επαγγελματία υγείας, του οικογενειακού γιατρού Φερρυπίν, εκείνου στον οποίο θα στραφεί ο γονέας για να ρωτήσει την ε, συμβουλή του για το αν θα πρέπει να εμβολιάσει το παιδί του κατά τη λαράς. Αυτός ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει να επιδείξει ηγετική στάση. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται ότι σε ορισμένες χώρες πολλοί είναι αυτοί οι επαγγελματίες υγείας που δεν επιδεικνύουν την στάση αυτή που θα έπρεπε και δεν παρακολουθούν και το εθνικό ημερολόγιο ή πρόγραμμα εμβολιασμών, πράγμα το οποίο μάλλον απαράδεκτο μου φαίνεται. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει οι επαγγελματίε υγεία σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπράξουν προ τον ίδιο στόχο και να μιλήσουν ξεκάθαρα για το φαινόμενο των κρουσμάτων Λαράς. Δεν χρειάζεται να μας στηρίζουν μόνο οι πολιτικοί, όπως δημοσίευσα την προηγούμενη εβδομάδα το άρθρο στο οποίο στους τους γιατρούς να αναλάβουν περισσότερο ενεργά μέτρα για την ε, ε, πρόοδο στους εμβολιασμούς. για συγκεκριμένες εκδηλώσεις που προβλέπονται και θα έχουμε και την σύνδρομη των ε, εμπειρογνωμίνων. Και κάθε φορά που κρίνει το κέντρο μας ότι υπάρχει μία απειλή, βλέπετε ότι ε, τότε στον ιστότοπό μας ε, δημοσιεύουμε μία έκθεση για θέματα υψηλού κινδύνου και θεωρούμε ότι οι υπεύθυνοι στον τομέα τους, της υγείας θα πρέπει να δώσουν συνέχεια. Επίσης, χρησιμοποιούμε και το Twitter και λαμβάνουμε μηνύματα από εσάς στο Twitter, ε, μηνύματα πολύ σύντομα, αλλά πολύ σημαντικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες από μολυσματικές ασθένειες, αλλά θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια ε, μικρόβια πρέπει να αντιμετωπιστούν, διότι δυστυχώς ανθίστανται στα φάρμακα. Και πιστεύω ότι το Κέντρο ε, Αντιμετώπισης Νόσων μπορεί να σας βοηθήσει όχι μόνο για το θέμα του AIDS, αλλά και για πολλά άλλα θέματα και ασθένειες. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την παρουσίαση αυτή Η Φρανσουά Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, η εισήγησή σας ήταν άκρος ενδιαφέρουσα για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα. Μιλήσατε για το θέμα της Ιλαράς και στη δική μου χώρα, στη Γαλλία, αντιμετωπίσουμε μεγάλο πρόβλημα για την αντιμετώπιση της ηλαράς, κάτι το οποίο είναι πονίδιστο, γιατί υπάρχει έλλειψη εμβολίων και υπάρχουν πολλοί επαΐοντες και οι δήμονες οι οποίοι δεν προτρέπουν τους γονείς να εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι απαράδεκτο γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στα σημερινά εμβόλια. Εδώ και 30-40 χρόνια υπήρχαν προβλήματα όπου θα, μπορούσαμε, θα μπορούσαν να υπάρξουν ανησυχίες ως προς τα εμβόλια. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι τα εμβόλια είναι άκρος κατάλληλα και δεν παρουσιάζουν κινδύνους για τα παιδιά. Μας είπατε λοιπόν ότι και εσείς προβάλλετε μία επικοινωνιακή πολιτική με τους υπεύθυνου υγείας. Αλλά θα έπρεπε να είμαστε πιο δραστήριοι και αυτό να ξεκινά από το Υπουργείο Υγείας για να προβάλλονται προγράμματα εμβολιασμού κατά της Ιλαράς, γιατί είναι απαράδεκτο στην Ευρώπη να έχουμε θανάτους από την Ιλαρά. Σήμερα έχουμε μία Ε, ειδική έκθεση για θέματα που αφορούν την αντίσταση στα μικρόβια με τον Πίτερ Λίζε. Έχουμε υποβάλει μία έκθεση και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορούμε να συγκρίνουμε τα δεδομένα με την κατάλληλη εποπτεία. Το σύστημα προειδοποίησης το δικό σας είναι πολύ σημαντικό και όταν υπάρχουν ε, συγκεκριμένα στελέχη που δείχνουν αυτή την, ότι επιτείνεται αυτή η αντίσταση, θα πρέπει να ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ ανθρώπου και ζώων. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το τρίτο θέμα. Δεν θα ήθελα να επανέλθω στον HIV, αλλά ως προς τη γρήπη. Φαίνεται ότι ε, ε, ε, επανερχόμαστε στο H5N1. Τι, πώς έχει κατάσταση σε σχέση με τα νέα εμβόλια, διότι ο, υπάρχει κίνδυνος, υφίσταται πραγματικός κίνδυνος και ποια είναι η θέση σας. Και ως προς την H5N1 ε, φαίνεται ότι αυτή η ασιατική γρήπη επανεμφανίζεται και αντιστέκεται σε κάθε μορφή αντιμετώπισης. Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ποια μέτρα προβλέπονται. Αυτό ήταν η πρώτη ερώτηση μέσα σε ένα φάσμα, η Λίντα Μακέβιν. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και που μας ε, μιλήσατε ε, επί της ουσίας ως προς την Ήλαρα είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε τα στοιχεία, γιατί βλέπουμε ότι οι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες ε, δυστυχώς έχουν, ε, ε, κατέχουν ένα ρόλο πρωταρχικό και βλέπουμε ότι δυστυχώς εξάγουμε και την ηλαρά σε τρίτες χώρες. Στη δική μου χώρα είχαμε να κάνουμε με έναν ανεύθυνο γιατρό και έναν ανεύθυνο δημοσιογράφο. Ο γιατρός ε, όμως ε, στην ουσία απομακρύνθηκε, αλλά πέρασε και το μήνυμα στους γονείς σε σχέση με τα εμβόλια. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την Ήλαρα αν έχετε τον αριθμό αναχώρα, ε, αριθμό κρουσμάτων αναχώρα. Θα ήθελα να μου αποσταλούν αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα για τη χώρα μου, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε προτεραιότητες, λοιπόν. Τι θα, πώς τις ορίζετε. Πώς είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα γιατί έχετε περιορισμένα μέσα. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στους ε, υπουργούς υγείας να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα ή στους γιατρούς. Ως προς τις προτεραιότητες, τις αιτήσιες προτεραιότητες σας, έχει μεγάλη σημασία η υγεία και για τους μετανάστες. Αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως κέντρο νόσων, δηλαδή κάτι που δεν κάνει κάποιος άλλος. Γιατί όταν μιλάμε εδώ για υγεία θέλουμε να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς και τι θα κάνουν στα κράτη. Γιατί διαφορετικά ε, κυνηγάμε την ουρά μας και η μεν και η δε. Εάν δεν μπορείτε λοιπόν να κάνετε τη διαφορά τότε αφήστε το σε κάποιον άλλο γιατί κάθε Μίκιο ασχολείται με θέματα υγείας και ισότητας, αλλά τι κάνει επί της ουσίας. Σε σχέση τώρα με την αντίσταση των ε, μικροβίων, θα ήθελα να μας πείτε τι κάνετε, γιατί έχουμε σωρία τροπολογιών όπου ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν τι κάνετε για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια στο δίνεκες. Επίσης μιλήσατε για ληστερία, για το e-coli, για γενικότερα δηλητηριάσεις από φαγητά. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, τι έγινε στη Γερμανία, γιατί εμεί μετά τα κρούσματα αυτά δεν ακούσαμε τίποτα άλλο. Ήθελα να ρωτήσω πώς συμμετείχατε εσείς στην αντιμετώπιση του e-coli. Νομίζω ότι θα σας υποβάλω και εγώ μία ερώτηση. Είδα ότι υπάρχουν γραμμές στον προϋπολογισμό για την ανάλυση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στις ασθένειες. Μπορείτε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο έπειτα. Όταν μιλάμε για μικρόβια, για ανθιστάμενα μικρόβια, Ίσως μιλάμε για θέματα που δεν είναι της απολύτου αρμοδιότητάς σας, αλλά να δούμε και το θέμα της ε, ευζοίας των ζώων σε σχέση με τα αντιστεκόμενα μικρόβια. Ίσως δεν είναι άμεσα στην εντολή σας, αλλά εάν υπάρχει, αν ασχοληθούμε με την ευζοία των ζώων, ίσως θα υπάρξει και μια αιτιώδη συνάφεια με ασθένειες σε επίπεδο ανθρώπου. Με την ΕΦΣΑ, με τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, είχαμε πολλές συγκρούσεις συμφερόντων. Και βεβαίως, αν κάνετε μία σύσταση για εμβολιασμό, αυτό έχει τεράστια επίπτωση ε, χρηματοδοτικής υφής. Μιλήσατε για την Γαλλία, για το Ηνωμένο Βασίλειο, για την Ιλαρά και πολλοί γιατροί ε, ζητούν να μην διενεργούνται εμβολιασμοί. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Πολλοί βεβαίως έχουν εμβολιαστεί και πολλά μικρά παιδιά έχουν μεγάλο πρόβλημα, προβλήματα με τον ύπνο επειδή ε, εμβολιάστηκαν. Πώς υπάρχει, πώς ορίζεται αυτή τη σχέση ε, κόστους ωφελίας. Ο καθηγητής Ζακ Σέρες είναι εδώ μαζί μας. Αν θέλετε κάτι να πείτε, εσείς μας εκπροσωπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορείτε να μας πείτε κι εσείς ε, ό,τι θα θέλετε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω κι εγώ το λόγο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ. Εγώ σας εκπροσωπώ εδώ και τέσσερα χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο και βλέπουμε ότι ο οργανισμός αυτός λειτουργεί πολύ καλά υπό τον πρώτο διευθυντή και υπό την, τον δεύτερο τώρα. Η, κυρία Μαλιόρη είναι εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να βρεθεί εδώ σήμερα, αλλά μιλώ και εξ ονόματός της. Έχει μεγάλη σημασία για μας να έχουμε μεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον για το κέντρο σας. Μιλήσατε για μία επίσκεψη υπό τον Γιώ Λάινεν, μίας αντιπροσωπείας και μιλάτε και για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η κυρία Γιανακούδάκη, η κυρία ε, Κάντενμπαχ, η κυρία Ροντ Μπέρεντ ζήτησαν να έχουμε κοινέ δραστηριότητες ή εκδηλώσεις. Αυτό είναι πολύ θετικό και μας οδηγεί στο ότι θα επανέλθουμε μαζί με την κυρία Μαλιόρη επί του θέματος, διότι στο παρελθόν δεν είχαν προβλεφθεί τέτοιες επισκέψεις. Κάναμε μια διαδικασία οικοτολογίας καθαρά στο παρελθόν, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η συζήτηση αυτή που προφέιτε Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Αυτό γενικά. Τώρα θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ το θέμα που έθιξε η κυρία Μακέβιν και η άλλη συνάδελφος για την Ιλαρά, για τα κρούσματα Ιλαράς. Έχει μεγάλη σημασία η αντιμετώπιση του θέματος και από το Κέντρο Ελέγχου Νόσων. Γιατί δεν θέλουμε να το δούμε à la Δηλαδή, οι μεγάλες χώρες θεωρούν ότι το κέντρο ελέγχου νόσων δεν θα πρέπει να ασχολείται με θέματα νοσολογίας. Γιατί εγώ είχα κάνει ορισμένα σχόλια όταν έκανε συστάσεις το κέντρο ελέγχου νόσων και πολλές χώρες και ιδιαίτερα οι τρεις μεγάλες είπαν όχι, δεν θέλουμε συστάσεις. Καταλαβαίνετε που μπορεί να οδηγήσει αυτό, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα εκεί όπου ανακύπτουν. Θα πρέπει λοιπόν να σας ε, ε, απασχολήσει και θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Γκροστέτ και Μακάβιν, γιατί βλέπουμε την ανάγκη μιας ε, εκβαθέων συζήτησης. Ιδιαίτερα οι μικρές χώρες είναι ιδιαίτερα είναι ευτυχείς, αλλά οι μεγαλύτερες χώρες αντιδρούν. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να μας απασχολήσει σε μια επικοινωνιακή πολιτική με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο που έχει έμεσα τεθεί επιτάπητος, δηλαδή η επικοινωνία με τους πολιτικούς, με το κοινό, τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Ένα παράδειγμα ήταν η γρήπη, η H5N1, όπου τα Εθνικά Κέντρα Υγείας ή τα Εθνικά Υπουργεία δεν μπορούσαν να ορίσουν επακριβώς την κατάσταση. Το θέμα αυτό καθοδηγήθηκε από, τα, από τους πολιτικούς, από τα μέσα, από κοινωνικούς φορείς που προέβαλαν κινήσεις οι οποίες δεν εντάσσονταν σε ένα ε, ρυθμιστικό πλαίσιο στον ΠΟΗ, στα Εθνικά Κέντρα Υγείας και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια επικοινωνιακή πολιτική. Είχαμε πολλά παραδείγματα, δηλαδή η αντίσταση των, ε, στα αντιβιωτικά είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Οι γιατροί συνταγογραφούν ακόμα και εκεί που δεν θα έπρεπε. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ε, χαίρομαι γιατί και αύριο θα μιλήσουμε για την αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιωτικά. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. γιατί ένα μικρό γατάκι όταν κάνει κάτι που δεν αρέσει στη μαμά, ε, η μαμά θα τήρει το ε, γατάκι, αλλά αν ένας γιατρός δεν πλύνει τα χέρια του, δεν απολυμανθεί ε, και ο ασθενής στη συνέχεια μετά από μία εβδομάδα αποβιώσει, τότε δεν, δεν μπορεί να συσταθεί αυτή η αιτιώδη συνάφεια. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι η επικοινωνιακή πολιτική σε θέματα υγείας που θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο. Γιατί ξέρουμε πολλά για, τις, για τους ιούς των νοσοκομείων, για τη μοριακή σύνθεση των ε, αντιβιωτικών, αλλά πολλές φορές συνταγογραφούν οι γιατροί εκεί που δεν χρειάζεται. Οι γιατροί, ας πούμε, δεν μπλένουν τα χέρια τους. Κάτι το πολύ απλό. Και τώρα, ε, ως προς το τελευταίο θέμα που αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, δημιουργήθηκε, είναι εξαιρετικός οργανισμός και διαθέτει μέσα. Το ΤΕΣΥ είναι το σύστημα εποπτείας που ε, στην ουσία ελέγχει τα επιμέρους στοιχεία. Γιατί παλαιότερα μόνο στη Στοκχόλμη βλέπαμε ότι αυτοί οι ασθενείς προέρχονταν από ένα μικρό χωριό. Γι' αυτό χρειάζεται ολοκληρωμένη εποπτεία και μετρήσιμη τρόπη εντοπισμού έτσι ώστε να ευεργεθούν περισσότερο όλοι από αυτό το μέσο, όχι μόνο για τις μολυσματικές ασθένειες, γιατί τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι ροές πληροφοριών θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε για χρόνιες ασθένειες ή για ασθένειες υψηλού κινδύνου. Αν δείτε το διαβήτη, ο διαβήτη μάλλον η διαφυτικοί, είναι πολύ πιο ευαλωτή σε μολυσματικές ασθένειες. Υπάρχει λοιπόν ε, αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ μολυσματικών ασθενειών και ορισμένων κατηγοριών ασθενών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε καλύτερη χρήση αυτών των μέσων, όπως το τέσι, που είναι το μέσον εποπτείας, δημιουργήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τομείς. Ξέρω ότι η εντολή σας ε, είναι περιορισμένη, το Συμβούλιο δεν σας επιτρέπει να επεκταθείτε, αλλά επειδή σας εκπροσωπώ, κάνω αυτή την έκκληση. Βρίσκομαι στο τέλος της δεύτερης θητείας μου και είμαι πεπισμένος ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη την εφαρμογή αυτού του μέσου και σε άλλους τομείς. Αυτή είναι μια συζήτηση η οποία θα ανακύψει φέτος ή του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και ε, χαίρομαι και με μεγάλη τιμή επιτελώ αυτό το έργο. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ που λάβατε το λόγο. Με μεγάλη ευχαρίστηση ε, ακούσαμε την εισήγησή σας. Αν θέλετε μπορείτε να αποστείλετε και μία επιστολή επί του θέματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σας δώσω το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ κυρία Γκροστέτ και κυρία Μακέβεν για τις ερωτήσεις που κάνατε για την Ιλαρά. Για να είμαι ειλικρινής και εγώ ντρέπομαι που εξάγουμε ασθένειες η Αμερική, ο Καναδάς, ε, η Λατινική η Αμερική. Ε, Ήταν περιοχές όπου δεν υπήρχαν κρούσματα Ιλαράς και τους τα φέραμε εμείς, ε, τα εξήγαμε εμείς. Ξέρετε για, για ποιον μιλάω, δεν μιλάω για τα κράτη-μέλη. Ε, Κάθε τέσσερις εβδομάδες δημοσιεύουμε μία ε, πολύ λεπτομερή ενημέρωση για τις χώρες ε, που δεν είναι ελεύθερες ηλαράς και με τα χαράς να σας διαβάσω το αρχείο. Ε, επίσης υπήρξε σύσταση από πλευράς του Συμβουλίου επί Ουγγρικής Προεδρίας σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών, αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύτηκε και ένα άρθρο μου, ε, όπου ε, ξεκάθαρα προκύπτει ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τους γιατρούς. Δηλαδή, όλο ένα και περισσότεροι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις αρμόδιες αρχές ε, της αλλά παρόλα αυτά εμπιστεύουν τον γιατρό τους. a very contagious ε, η κάλυψη με τα εμβόλια φτάνει το 95% και λειτουργούν καλά τα εμβόλια. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά φανταστείτε να υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν θέλουν να δραστηριοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί η νόσος. Οι γονείς δεν είναι πεπισμένοι, για να το πω με απλά λόγια, ότι πρέπει να ακολουθήσουν το, πολιτικό, ε, το εθνικό πρόγραμμα ε, ανοσοποίησης, το οποίο είναι και δωρεάν. Οπότε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα κρούσματα ελαράς. Ε, ε, ορισμένοι υποτιμούν και τη σημασία της νόσου. Ναι, μεν, αλλά 25% των τωρινών ε, κρούσματων ε, οδηγούν σε πνευμονία και άρα πρέπει να νοσηλευθεί ο ασθενής και μία στα χίλια μπορεί να προκύψει και εγκεφαλίτιδα, πάρε εγκεφαλίτιδα μάλλον. Οπότε καταλαβαίνετε δεν πρέπει να υποτιμούμε την ασθένεια και με τέτοια συμπεριφορά του κοινού δύσκολα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους. Ε, ξέρετε τι κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης. Επίσης, από πλευρά κοινωνικών επιστημών μελετούμε τρόπου με τους οποίους θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των ε, πολιτών αλλά και των επαγγελματιών του τομέα υγείας ε, καθώς και να υιοθετήσουμε μια περιφερειακή προσέγγιση με ένα ε, κουτί εργαλείων αν θέλετε για μεμονωμένε περιστάσει. γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία λύση. Επίση, ένα πακέτο και το ε, ενημερωτικό το οποίο θα δημοσιεύσουμε του χρόνου. Δύσκολα μπορούμε να καταμετρήσουμε όμως τα αποτελέσματα γιατί φυσικά αν αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμών θα μειωθεί ο αριθμός των ε, κρουσμάτων. Επίσης υπάρχουν οι λεγόμενες catch-up ε, εκστρατείες ε, για τον εμβολιασμό μικρών παιδιών ενός δύο χρονών γιατί χρειάζεται και η επαναληπτική, το επαναληπτικό το εμβόλιο και ορισμένες χώρες δεν, έχουν, δεν δραστηριοποιούνται για αυτό το επαναληπτικό εμβόλιο. Αυτές είναι οι εκστρατείες ε, catch-up. Τώρα, Πιστεύω ότι έχουμε τα στοιχεία, αναφερθήκατε κι εσείς στα ε, στοιχεία που έχει το κέντρο μας. Ε, έχουμε το EARSNET, δηλαδή ένα δίκτυο εποπτείας ε, που έχει ιδρύσει το κέντρο μας και πριν από τρεις εβδομάδες πήγα στη μεγαλύτερη διάσκεψη, ονομάζεται ICA στο Σικάγο για τις μεταδιδόμενες ασθένειες και ένας από τους ο Καθηγητή Λίβαμορ από το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι από του επιφανέστερού ειδικού στην αντιμικροβιολογική μελέτη χρησιμοποίησε, ξέρετε, ε, στοιχεία από το κέντρο μας, ε, τρόπους ε, μέτρησης της μικροβιολογικής αντίστασης. Επίσης, μου ζητούνται τα στοιχεία του κέντρου μας για χρήση σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε προώρα να δούμε τις ε, αλλαγές ε, στις τάσεις και να αντιδράσουμε. Επίσης θυμηθείτε τον ιό, το στέλεχος του ιού του Νέου Δελχή. Κάναμε την έκθεση αξιολόγησης πριν από ένα χρόνο και μπορώ να σας πω ότι δεν είναι καθόλου καλή η κατάσταση. Έχουμε ε, κάνει και διάφορε αξιολογίες για το λεγόμενο CPE και προσπαθούμε και πάλι να πείσουμε του επαγγελματίε ε, του κλάδου ότι πρέπει να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή για τέτοιε θεραπευτικές αγωγέ, όπως είπε και ο καθηγητής Χίρης ε, αλλά ε, βοή εν είναι δυστυχώς προς το παρόν. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πορό θα ξεκινήσει μια δική της εκστρατεία. Έχουμε ε, εργαλεία στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε την αντιμικροβιολογική αντίσταση για τη γρήπη. Είδαμε ένα ανακοινωθέν τύπου για το H1N1 από τον ΦΑΟ. Ναι, υπάρχουν ανησυχίες για κάποιες μεταλλάξεις του ιού. Κάναμε μια ταχύτατη ε, ε, αποτίμηση κινδύνου και από δική μας πλευράς και μετά από διαβούλευση με την ΠΟΗ κρίνουμε ότι δεν, δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος, παραμένει στα ίδια επίπεδα ο κίνδυνος, ε, πλην όμως θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις νέες μεταλλάξεις αυτού του στελέχους του ιού H1N1 και παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις, ε, κυρίως ε, στο στον τομέα της ε, γεωργίας. Ξέρετε, ανάμεσα στο Χόλμη και τις Βρυξέλλες υπάρχει πολύ καλή σύνδεση και ήρθε ένα κλιμάκιο από την φαρμακοβιομηχανία στο κέντρο μας για να συζητήσουμε τα το θέμα της γρήπης, το νέο εμβόλιο για την επερχόμενη σεζόν. Κάναμε μια ανοιχτή συζήτηση και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία ανησυχίας. Τα εμβόλια είναι υψηλής ποιότητας. Επίσης ε, συζητήσαμε, διερευνήσαμε νέους τρόπους ε, μελλοντικής συνεργασίας και αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης, ε, θυμάστε τις συζητήσεις που έγιναν για την εκλαμψία πριν από ένα χρόνο ε, όχι μόνο για τον κίνδυνο της ναρκοληψίας ε, αλλά διότι είναι ένα θέμα που μπορεί να υποσκάψει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε σχέση με ένα εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Και για να είμαι ειλικρανής, ε, αυτό το όλο θέμα τη ηλαρά ε, έχει τόση σημασία λόγω όλη αυτή της συζήτηση περί αυτισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, άλλων νόσων που μπορεί να συνδέονται με τον παιδικό εμβολιασμό. Χωρί όμω να υπάρχει καμία ουσιαστική αιτία. Για την αρκοληψία λοιπόν αρχίσαμε μια ευρύτατη ε, μελέτη στην Ευρώπη. Πάνω από 100.000 ε, παιδιά εξετάστηκαν. Ε, διαθέσαμε πολλά κονδύλια για αυτή τη μελέτη και αναμένουμε τα πορίσματα. Το φθινόπωρο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα. Αλλά μπορούμε να αναμένουμε κάποια χρήσιμα αποτελέσματα το φθινόπωρο Τι άλλο. Για το ΙΧΑΚ, το e Πολλοί ε, ε, συζητούν το θέμα των ανισοτήτων ε, στον τομέα της υγείας και πολλές από αυτές τις συζητήσεις, πώς θα το έλεγα, γίνονται σε γενικότερο επίπεδο. Εμείς πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, πώς να ενημερώσουμε για τις μολυσματικές ασθένειες. Δείτε τη φυματίωση. Εκεί υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, διότι οι έχοντες ποτέ δεν προσβάλλονται από τη φυματίωση. Η φυματίωση λοιπόν είναι κατεξοχήν ο τομέας των αν ισοτήτων στον τομέα της υγείας και όλα τα κρούσματα είναι σε μία χώρα μόνο ή τουλάχιστον το 90% είναι σε πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε ποια είναι αυτά τα κράτη-μέλη, ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά σε κάποιες χώρες, δεν θα κατονομάσω καμία χώρα, αλλά αυτά τα παιδιά πρώτον ε, δεν, ε, ε, δεν έχουν ούτε τη σωστή διάγνωση, ούτε έγκυρη διάγνωση, ούτε και σωστά φάρμακα, δηλαδή φάρμακα κατάλληλα για παιδιά παιδιά. Ε, πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την καταπολέμηση της φυματίωσης διότι αυτή η νόσος ε, είναι η κατεξοχή νόσος ε, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Τώρα εμβολιασμός για την ε, φυματίωση. Κοιτάξτε, όσοι εμβολιάζονται είναι μάλλον ε, καλλιεργημένοι άνθρωποι που αποφασίζουν τέλο πάντων να μην εμβολιαστούν. Εντάξει, η επιλογή του είναι. Αλλά ε, από την άλλη πλευρά έχουμε και τι ευάλωτε πληθυσμιακέ ομάδε και αυτό μελετούμε. Πώ μπορούμε να φτάσουμε σε αυτού του ανθρώπου που θέλουν να εμβολιαστούν αλλά δεν έχουν δυνατότητα να προμηθευτούν εμβόλιο. Ένα άλλο παράδειγμα και αναφερθήκατε κι εσεί αυτό είναι ο ιό HIV και χαίρομαι πολύ που το συνδέσατε με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των ιών διότι εάν δεν ε, διαγνωστεί εγκαίρος και πρόωρα ο ιός, αν δεν κατοχυρώζεται πρόσβαση στη θεραπευτική αγωγή, πάλι σημαίνονται ανισότητα ε, τέλος. Οι χώρες ε, Ε, και ε, οι γυναίκες ε, κυρίως που δεν κάνουν το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου βρίσκονται στις φτωχότερες χώρες και πάλι εδώ έχουμε θέμα ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Ξέρετε δεν είναι και πυρηνική φυσική, είναι εύκολο εάν έχουμε την απαιτούμενη δέσμευση και αν πείσουμε τις κυβερνήσεις ότι πρέπει να δώσουν σημασία σε αυτό το θέμα για το η κόλλη ήταν το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αιστεία μόλυνσης από αυτό το στέλεχος του E. στην Ευρώπη. Πολλοί μολύνθηκαν στην Γερμανία. Ε, και πολλοί γιατροί εντυπωσιάστηκαν από τις ε, ε, αρνητικές επιπτώσεις αυτής της νόσου. Ποτέ δεν είχαν δει τόσο σοβαρές περιπλοκές και ο ρόλος του κέντρου μας ποιος ήταν δώσαμε ορισμούς για, τα, για συγκεκριμένα κρούσματα, δώσαμε την καθοδήγηση για συναφή ζητήματα, διότι ήταν σπάνιο αυτό το στέλεχος και τα εργαστηρία δεν ήταν έτοιμα να αντιμετωπίσουν ε, τέτοια στελέχη και άρα τα καθοδηγήσαμε επίσης επιστημονικά δεδομένα. Τώρα ξέρουμε ότι αυτή η επιδημία περιορίστηκε κυρίως στη Γερμανία παρότι εμφανίστηκαν και κάποια κρούσματα στη Γαλλία. Στην αρχή όμως δεν το ξέραμε αυτό προφανέστατα και άρα θέλαμε να συλλέξουμε δεδομένα από όλες ε, τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα εισαγάγουμε στο σύστημα σύστημά μας. Κινητοποιήσαμε επίσης ε, το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων για τις ε, ασθένειες που μεταδίδονται από τον αέρα ή μέσα από το νερό και οι ειδικοί λοιπόν για κλινικές περιπτώσεις μας συμβούλευσαν για την αντιμετώπιση αυτών των τόσο πολυάριθμων κρουσμάτων και καθώς και για την νοσηλευτική τους αγωγή. Συνεργαζόμαστε επίσης με το Ινστιτούτο Ροχανκούν και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά ε, φυσικά συνεργαζόμαστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας ε, Τροφίμων και τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και έτσι καταλήξαμε σε διάφορα συγκεκριμένα μέτρα που κρίνουμε ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Ποια διδάγματα μπορούμε να αντιλήσουμε τώρα από αυτήν την επιδημία. Αυτές οι επιδημίες μπορούν να σημειωθούν σε πολύ καλά εξοπλισμένες σε εισαγωγικά χώρες, οπότε προσοχή να έχουμε όλη επίγνωση το ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Οπουδήποτε δεν μιλάμε μόνο για μια φτωχή χώρα που δεν έχει τους απαιτούμενους πόρους, μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Προσοχή λοιπόν. Επίσης, ξέραμε ότι υπήρξε καθυστέρηση ως προς την κοινοποίηση. Την περασμένη φορά που ήμουν εδώ, κάναμε τη συζήτηση για την υπατήτηδα και ξαφνικά η κυρία Ντάκμαρον Μπέρεντε με ρώτησε Ε, μου έκανε ερωτήσει για την ε, επιδημία στην ε, Γερμανία και ξέρουμε ότι υπήρξε καθυστέρηση 21, 21 ημέρες, δηλαδή καθυστέρησε η όλη διαδικασία ενημέρωσης για να περάσουν πληροφορίες από τους γιατρούς σε ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία το Ινστιτούτο Περκόχ δηλαδή πήρε το σήμα με μεγάλη καθυστέρηση ενώ ε, σε εθνικό επίπεδο, ενώ εμείς μπορέσαμε κατευθείαν να εισαγάγουμε τις πληροφορίες στο σύστημα. Ξέρετε, σε, επιμέρου στις επιμέρους χώρους έχετε διάφορα επίπεδα ο γιατρός, το τοπικό επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο, μέχρι να φτάσει η πληροφορία στο κεντρικό επίπεδο. Και παρότι έχουμε εξαιρετικά συστήματα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, λειτουργούν πάντα τα συστήματα. Προσοχή και σε αυτό λοιπόν. Ξέρουμε επίσης ότι οι επαγγελματίες του κλάδου, οι γιατροί πρέπει να προσέξουν γιατί έχουν ιδιαίτερο ρόλο και κατακλείζονται από το μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και δεν λειτουργούν πάντοτε σωστά. Σχετικά με τη διάσκεψη του ΟΗΕ για τις κλιματικές αλλαγές, επίσης χαίρομαι που το αναφέρατε και εμείς ε, διοχετεύουμε πολλά κονδύλια για αυτό το θέμα. Ε, ξέρετε ότι έχουμε και τα, τα τίξ, ε, τα τσιμπούρια, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε στη Σουηδία που μεταδίδουν ασθενείες και, και η μεγάλη αύξηση του αριθμού των τσιμπουριών ε, μπορεί αυτό να οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές στην Ελλάδα αλλά όχι μόνο και στην Ιταλία έχουν σημειωθεί κρούσματα ελονοσίας που μπορεί να συνδέονται με αυτές τις κλιματικές αλλαγές και έτσι κάνουμε έρευνες για να δούμε οι κλιματικές αλλαγές σε ποια σχέση έχουν με την εμφάνιση ε, ε, νέων κρουσμάτων σε αυτές τις μεταδιδόμενες ασθένειες και διοχετεύουμε κονδύλια. Ξέρετε δεν είναι και πολύ δημοφιλές το θέμα και πάντοτε εγώ προσωπικά ανησυχώ διότι από πλευράς δημόσιας υγείας, από ιατρικής πλευράς ε, ανησυχώ ότι δεν αποδίδεται ε, το βάρος ε, σε αυτό το θέμα. Θεωρούν όλοι ότι είναι ένα περιβαλλοντικό ζήτημα οι κλιματικές αλλαγές αλλά κρούω τον κόδωνα του κινδύνου γιατί οι κλιματικές αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν σοβαρότατα τη δημόσια υγεία. Ο κύριος Λάιτερ, ευχαριστώ. Νομίζω απαντήσατε όλες τις ερωτήσεις εκτός από μία αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Για αυτά τα τσιμπούρια είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι από το αρχιπέλαγο ε, και, ε, και η μπορέλια και η φυματίωση μεταδίδονται μέσα από τα τσιμπούρια και είναι δύο σοβαρότατες μεταδοτικές ε, ασθένειες. Α, ναι, ξέχασα, λέει ο κύριο Πρέγκερ, τα περισύγκρου συμφερόντων. θα, τα, θα απαντήσω. Έχουμε λοιπόν στον οργανισμό μας ότι ε, ε, ε, έχουμε στον οργανισμό μας εμπειρογνώμους που ασχολούνται με αυτό το θέμα που ιδιαίτερη σημασία σε αυτό και γίνονται αξιολογήσεις κίνδυνο από τους δικούς μας ειδικού. Πέρσι το Διοικητικό μας Συμβούλιο υιοθέτησε μια πολιτική για τη σύγκρουση συμφερόντων, αλλά υπήρξε ένα κόλλημα. Ε, έπρεπε να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση γιατί μας το ζήτησε ο, Ευρωπαϊκός, ο Ευρωπαίος Αρμόδιος για τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ή μας έκαναν κάποιες ερωτήσεις, απαντήσαμε μετά κάποιες άλλες ερωτήσεις και περιμένουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Ταυτόχρονα Πήγαμε στην ομάδα εργασία τη DG Sanko για το θέμα της σύγκρουση των συμφερόντων και θα θεσπίσουμε δική μας πολιτική κυρίως για τη γρήπη. Ε, ε, Διαβολευόμαστε με όλους. Μάλλον, ζητούμε από τα μέλη του προσωπικού μας να ε, αναρτήσουν στην ιστοσελίδα μας τα πάντα περί σύγκρουσης ε, συμφερόντων. Έγινε αυτό. Υπάρχουν τα στοιχεία ε, στην ιστοσελίδα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Περιμένουμε τη γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαίου αρμοδίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και υπάρχει και το θέμα Ε, της ε, κατοχής ομολογιών σε επιχειρήσεις κτλ. Μάλιστα λέει ο κύριος ε, Σλάιντερ, ευχαριστούμε και είμαι σίγουρος ότι αν προκύψουν άλλα επιδημιολογικά προβλήματα του χρόνου θα τα αντιμετωπίσετε με την ίδια σοβαρότητα που και αυτά που μας περιγράψατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι και το τελευταίο σημείο της ημερής διάταξη διάταξης αύριο και μην ξεχάσετε και τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίες και ελάτε εγκαίρως γιατί μπορεί μία μέρα, δεν ξέρετε ποτέ, να αρχίσουμε και εγκαίρως.